Καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες ε, της Επιτροπής μας με κάποια μικρή ε, καθυστέρηση. Η αλλαγή της εθούσης φαίνεται ότι δημιούργησε κάποια προβληματάκια. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πάρα πολύ σύντομες ε, πριν ξεκινήσουμε τις κανονικές εργασίες της Επιτροπής μας. Η πρώτη ανακοίνωση είναι ότι έχει ακυρωθεί η ε, συνεδρίαση της Πέμπτης το απόγευμα. Δεν θα συνεδριάσουμε λοιπόν Πέμπτη απόγευμα. Επίσης, σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως σχετικά με το feedback όσον αφορά ε, τον τριμερή διάλογο που έγινε μέχρι προχτές ε, το βράδυ και μάλιστα έφτασε και πολύ αργά, είναι ένα σημείο το οποίο διαγράφεται ε, δεν υπήρξε ε, οποιοδήποτε συγκεκριμένο, οποιαδήποτε συγκεκριμένη έκβαση από τον τριμερή αυτό διάλογο, επομένως δεν έχει έννοια αυτή η ενημέρωση. Έχετε κάποιο πρόβλημα, ρωτάει η Πρόεδρος. Όχι, συνεχίζουμε λοιπόν. Τρίτο σημείο που θέλω να σας δείξω. Σήμερα δυστυχώς το πρωί δεν έχουμε διερμηνία προς όλες τις γλώσσες λαμβάνοντας υπόψη ε, επίσης ότι, κυρίως μάλλον, ότι η αίθουσα αυτή δεν έχει όλες τις απαραίτητες ε, καμπίνες, αλλά το πρόβλημα αυτό θα το ξεπεράσουμε διότι σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί θα ξαναβρούμε τη συνηθισμένη μας ε, αίθουσα στην πλευρά του κτηρίου Γιάννα που έχει όλες τις καμπίνες που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν κάποιος θέλει να σχολιάσει, να αντιδράσει ε, στα όσα είπα μέχρι τώρα. Αν όχι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη έτσι όπως την έχουμε προβλέψει. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 4, ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Η Μαρίτα Ούτσκοφ είναι η εισηγήτρια. Θα δώσω στην εισηγήτρια το λόγο και θα συνεχίσω με τους σκιώδεις και με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα θελήσουν να πάρουν το λόγο. Μαρίτα. 400 ehm, Έχουμε πάρει περίπου 400 τροπολογίες για τον κανονισμό αυτό, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ταυτοποίησης και εμπιστοσύνη. Από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, οι διαφορές απόψεων δεν είναι τόσο μεγάλες. Οπότε υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με ένα κείμενο που θα είναι γενικά αποδεκτό. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με το τμήμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κανονισμού και μετά να εξετάσουμε τα θέματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Γενικά θα μπορούσα να σας πω ότι η πρόκληση είναι τώρα να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο ευθυγραμμίζεται με το τμήμα του κανονισμού για το οποίο έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Ξέρω ότι υπήρξε η ανάγκη να χωρίσουμε το κείμενο στα δύο μεταξύ των δύο επιτροπών. Αλλά το νομοθετικό κείμενο είναι έτσι συντεταγμένο ώστε να είναι πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία διαχωρισμού. Αν αλλάξουμε ένα άρθρο, τότε όλο το πλαίσιο τροποποιείται. Είναι σημαντικό λοιπόν <clears throat> και για μένα και για τους κοιόδης εισηγητές να μπορέσουμε να συντονίσουμε λίγο καλύτερα μέσα στην με τον κύριο Γκάλο, τον ε, εισηγητή της Επιτροπής ΙΜΚΟ, το κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε. Για τις τροπολογίες αυτές καθεαυτές, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι να πω κάτι σε επίπεδο αρχών, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Το πρώτο σημείο που πρέπει να μας ε, απασχολήσει είναι η έννοια της αυθεντικοποίησης έναντι της αναγνώρισης. Έχουμε τις, ταυτότητες, ε, τροπολογίες που προσπαθούν <clears throat> να ε, καθορίσουν τι ακριβώς θα πρέπει να είναι η ταυτοποίηση από το σύστημα ή η αυθεντικοποίηση. Δηλαδή ότι μόνο τα στοιχεία αυτά που είναι απαραίτητα για αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να αποκαλύπτονται κατά τη διαδικασία αυτή. Επομένως <clears throat> δεν θα πρέπει να δίδουμε υπερβολικά πολλά στοιχεία πληροφοριακά στο σύστημα αυτό. Η, η άποψή μου είναι ότι βέβαια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποκαλυπτονται κατα τη διαδικασια αυτη επομενως δεν θα πρεπει να διδουμε υπερβολικα πολλα στοιχεια πληροφοριακα στο συστημα αυτο η αποψη μου ειναι οτι βεβαια καθε κρατος μελος θα πρεπει να ειναι σε θέση να θεσπίσει τη δική του δομή, τη δική του αρχιτεκτονική για τη διαδικασία αυτή ταυτοποίησης. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να λειτουργεί αυτό το σύστημα και με τα εθνικά συστήματα και με το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν μια δομή η οποία έχει αρνητικές διακρίσεις εναντί των χωρών που θέλουν να διατηρήσουν τα εθνικά του συστήματα τα οποία δεν βασίζονται στην αναγνώριση τόσο πολύ όσο στην ταυτοποίηση. Που χρησιμοποιούν λοιπόν <clears throat> μία πιο απλή μέθοδο για να αναγνωρίζουν ή να ταυτοποιούν τους χρήστες. Εγώ θα παραμείνω σε αυτά τα οποία είπα προηγουμένως σε σχέση με τα αμοιβαία πρότυπα για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην τεχνολογική του ουδετερότητα, ώστε τα κρατημέλη να έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν τα πλαίσια τους. Ένα δεύτερο σημείο είναι τώρα η υποστασία δεδομένων. Το άρθρο 11 του κανονισμού καλύπτει μόνο τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Αλλά υπάρχει κάποια ανησυχία σε σχέση με τα θέματα αυτά. Και αυτό αφορά και το τμήμα του κειμένου που έχει να κάνει με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Παραγωγή χάρη τους μηχανισμούς επαλήθευσης που πρέπει να υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος για να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό. Είναι επαρκή οι γενικέ ε, ρυθμίσει για την προστασία των δεδομένων ή πρέπει σε αυτή την περίπτωση να θεσπίσουμε και περαιτέρω προδιαγραφές και διατάξεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να ενισχυθούν οι πρόνοιες για την προστασία των δεδομένων. Το σημείο 3 επίσης είναι πολύ σημαντικό. Το να δώσουμε προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα για ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαμεθοριακού χαρακτήρα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η Κομισιόν δεν έχει καθορίσει κάποια ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας. Τι ακριβώς πρέπει να αναπτυχθεί πρώτα και να εφαρμοστεί. Θέλουμε να συνδέσουμε τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτότητας των διαφόρων κρατών μελών, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η Κομισιόν και τα κατημέλη να εστιάσουν σε διαλειτουργικότητα για αυτές τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χαρακτήρα που έχουν τη μεγαλύτερη εμβέλεια σε διαμεθοριακό χαρακτήρα και έχουμε καταθέσει τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ένα ερώτημα το οποίο παραμένει και το οποίο πρέπει να διαλευκάνουμε επί τη βάση των τροπολογιών είναι το κατά πόσο όλες οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό είναι πράγματι απαραίτητες. Παραδείγματος χάρη, η επαλήθευση ταυτότητας σε μία σελίδα εισόδου. Για κάθε όμως μορφή υπηρεσίας εμπιστοσύνης θα πρέπει να συζητήσω με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε κατά πόσο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην νομοθεσία, στον κανονισμό αυτό. Πρέπει καταρχήν να γνωρίσουμε ποιες είναι οι συνέπειες των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα υιοθετήσουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε νομοθεσία η οποία θα είναι τροχοπέδη για περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη. Πέμπτο και τελευταίο σημείο. Η κατεχώρηση και οι εκτελεστικές πράξεις. Αυτό είναι ένα θέμα φυσικά οριζόντιου χαρακτήρα και είναι πολλές οι ρήτρε στο σχέδιο κανονισμού που μεταφέρουν εξουσίες στην Κομισιόν για να εφαρμόσει για να ε, εγκρίνει εφαρμοστικές, ε, μάλλον εκτελεστικές ή κατεχώρηση πράξεις. Και εδώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Υπάρχουν ορισμένα μέλη που βλέπουν με, με πολύ σκεπτικισμό την ιδιαίτερη εξάρτηση από τις κατεχώρηση πράξεις. Δεν έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά ε, πλήρως, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για αυτά. Ευχαριστώ πολύ Μαρίτα. <clears throat> Ξέρω ότι έχεις κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Υπάρχουν ε, πάνω από 449 τροπολογίες ε, και επομένως πολλή δουλειά ε, έχουμε ακόμα. Πιλάρντερ Καστίγιο, πρώτη σκιώδη συγγήτρια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μεταξύ των άλλων έχει σημαντικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς της εσωτερικής ψηφιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας από τους αδιαμφισβήτητους στόχους που είναι και μια υψηλή προτεραιότητα για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το ανοιχτό πνεύμα που κράτησε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν επιτυχή, υπήρξε μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των στοιχειωδών εισηγητών παρά τις αναπόφευκτες διαφορές απόψεων μεταξύ τους, νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο. Τουλάχιστον από την πλευρά της Επιτροπής μας, τη ΣΥΤΡΕ. Θα σταθώ τώρα σε ορισμένες τροπολογίες. Κάποιες τροπολογίες δηλαδή που έχω παρουσιάσει εγώ όπως και οι συναδελφοί μου. Είναι γεγονός ότι η συζήτηση για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης είναι πιο προχωρημένη. Αλλά αυτό είναι ένα από, όχι το μοναδικό θέμα, είναι ένα από τα θέματα στα οποία έχω επιμείνει περισσότερο με τις τροπολογίες μου και αυτό θέλω να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κάποια δυσκολία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον διαφορετικό ορισμό που δίδονται στους παρόχους υπηρεσιών ε, εμπιστοσύνης και τους διακεκριμένους κατά κάποιο τρόπο παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Δεν ξέρουμε πώς η ρυθμιστική αρχή θα μπορέσει να εφαρμόσει τον έλεγχο αυτό που αναφέρει το άρθρο 13 του κειμένου της Κομισιόν, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η, ένας κατάλογος παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και δεν υπάρχει και μια διαδικασία με την οποία αυτοί θα ανακοινώσουν και θα κοινοποιήσουν την δραστηριότητά του. Πώ μπορεί να γίνει αυτό αν δεν υπάρχει διαδικασία για να κοινοποιείται αυτή η δραστηριότητα στι ρυθμιστικέ αρχέ. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία πρόταση για να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το σύστημα αυτό. Και η τροπολογία 278 που έχει παρουσιαστεί από ένα συναδελφό μας, τον Σαΐτ Καρίν, στο άρθρο 15.1, που ζητά να υπάρξει μια πιστοποίηση για τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Ένα δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός μέσα σε εισαγωγικά οικοσυστήματος εμπιστοσύνης για να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ψηφιακή οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι η πιστοποιημένοι ε, πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνη θα είναι πιο εύκολο να παρέχουν τι υπηρεσίε του. Το άρθρο 17 επιτρέπει αυτοί οι πάροχοι να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσιών από τη στιγμή που έχουν κοινοποιήσει στον αρμόδιο εποπτικό φορέα την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε αυτή τη δραστηριότητα ακόμα και αν αυτός ο αρμόδιος φορέας δεν έχει επαληθεύσει τα στοιχεία τους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκ των υστέρων προβλήματα όμως και θα μου φαινόταν πιο λογικό το να μην μπαίνουν σε αυτόν τον κατάλογο των πιστοποιημένων παρόχων μέχρι ότου οι αρμόδιοι φορείς έχουν κάνει την επαλήθευση των στοιχείων αυτών των πορέων. Αυτά αναφέρονται στις τροπολογίες 323, 324, 322, 23, 24. Υπάρχουν όμως άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει με διαφορετικές τροπολογίες τα θέματα αυτά και έχουν παρουσιάσει προτάσεις οι οποίες και αυτές είναι ενδιαφέρουσες. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που να συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο όλων των τροπολογιών και που είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους. Τέλος, όταν πρόκειται για αυτό που λέει το άρθρο 10, τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ δεν αναφέρεται αν πρέπει να βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και επίσης δεν αναφέρεται ποιος είναι αρμόδιος για να επαληθεύσει το κατά πόσο συνάδουν τα χαρακτηριστικά τους με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πόσο λοιπόν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες με άλλες χώρες, ευρωπαϊκές ή με άλλες χώρες και πώς θα γίνει η επαλήθευση των παρόχων αυτών. Εδώ έχουμε λοιπόν την τροπολογία 223 που επιφορτίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το να προβεί στην ε, επαλήθευση αυτών των ε, συμφωνιών με τρίτες χώρες. Αυτό μου φαίνεται μια πολύ καλή ρύθμιση. Τώρα υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία δεν προφθαίνω να τα διεξέλθω. Παραδείγματο χάρη η ανάγκη να υπάρξει αυτή η ουδετερότητα σε τεχνολογικό επίπεδο που είναι στην τροπολογία 146 και 63 η επίση ανάγκη διαβούλευσης με τον ιδιωτικό τομέα προτού εγκριθούν οι μελλοντικέ ε, κατεξουσιοδότηση τα κτλ. Υπάρχουν τροπολογίε όπως οι 473, 475, 93 αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ότι είμαι απόλυτα διατεθειμένη να προχωρήσω σε διάλογο και σε συνεργασία με όλους τους κοιόντες εισηγητές. Νομίζω πράγματι ότι μπορούμε ως Επιτροπή Ήτρε να συμβάλλουμε στο να υπάρξει ένα καλό έγγραφο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πυράλντερ Καστίγιο. Ο κύριος Κρόιτσμαν από την Άλντε Σκιώδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. από τις τροπολογίες είναι φανερό ότι χρειάζεται σε πολλά σημεία να υπάρξει επανεπεξεργασία του κειμένου της Κομισιόν. Είναι πολλές φορές πολύπλοκο το θέμα αυτό και με πολλές λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογίες σε διάφορα σημεία. Θα αναφερθώ σε μερικές από τις πιο σημαντικές. Καταρχήν το κεφάλαιο EID, η ηλεκτρονική υπογραφή. Εδώ θα πρέπει πάντα η επαλήθευση ταυτότητας να γίνεται με ένα τρόπο ο οποίος δεν έχει αμφισημίες και παραγωγός χάρη σε περιπτώσεις όπου πρέπει να υπάρξει μια επαλήθευση ηλικίας για τους χρήστες. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται και επιτρέπονται από τα εθνικά συστήματα. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν αν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να τροποποιηθούν τα συστήματα αυτά και να εναρμονιστούν. Έχουμε προτείνει επίσης τροπολογίες που αφορούν την ε, πρόσβαση σε διαμεθοριακές υπηρεσίες. Και εδώ πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Δεν θα είναι δυνατόν τα συστήματα τα εθνικά να επιτρέπουν πρόσβαση σε άλλες χώρες με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που ισχύει στις χώρες αυτές. Επίσης θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να συγκρίνουμε τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επαλήθευσης ε, ταυτότητας και υπάρχουν τέτοια πιλωτικά προγράμματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη συσσωρευμένη εμπειρία για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να παρέμβουμε ιδιαίτερα στην αγορά γιατί προχωρά η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα αυτό και πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη. Δεν πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να νομοθετήσουμε υπερβολικά στον τομέα αυτό. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θέματα της αστικής ευθύνης. Όταν έχουμε υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται επιστοποιημένες θα πρέπει να υπάρχει ένα υψηλότερο βέβαια επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με τους παρόχους από τρίτες χώρες δεν πρέπει να εμποδίσουμε το να δίδουν τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπόκειται σε υπερβολικές ε, υποχρεώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν και οι πολίτες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Και φυσικά πρέπει να υπάρξει μια αρχή εποπτική σε ό,τι αφορά αυτές τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Πριν αρχίσει την ε, δραστηριότητά του ένας, ε, ένας πάροχος υπηρεσίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ε, προϋποθέσεις και όχι μόνο μετά από έξι μήνες. Τέλος, Έχουμε πάρα πολλή εργασία γιατί υπάρχει και το θέμα της ε, κατανομής αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Κατά την άποψή μου, οι θέσεις των μελών της Επιτροπής ΙΤΡΕ δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα μεταξύ τους και μπορούμε να καταλήξουμε σε λογικές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ehm, Σας ευχαριστώ. Ε, από τους Πρασίνους. Η κυρία Νεστόιτερ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους με τους οποίους εργαστήκαμε για αυτήν την έκθεση. Building trust, οικοδόμηση εμπιστοσύνη είναι οι δύο πρώτε λέξει τη οδηγία και αυτό θα πρέπει να είναι και ο πρώτο μα στόχο. Ε, με χαρά βλέπω ότι υπάρχουν ε, ε, ε, ιδέες ε, κατά αυτή την έννοια οι οποίες δεν είναι μόνο μου αλλά είναι και των εκπροσώπων των άλλων πολιτικών ομάδων. Ε, είναι ουσιώδου σημασίας και θα πρέπει να αποτελέσουν το κέντρο της, των προτεραιοτήτων μας. Είναι πολύ θετικό το ότι συνεργαστήκαμε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα σε πάρα πολύ καλό πνεύμα. Νομίζω ότι η ταυτοποίηση δεν αφορά την τεχνική μη εναρμονισμένη μεταξύ των μελών, κρατών μελών διαδικασία. Κατά την άποψή μου είναι ε, όλες αυτές ε, οι διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας που δεν έχουν ε, ομοιογενοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχει ένα τεχνικό σύστημα ε, και η κάθε χώρα έχει βρει διαφορετικές λύσεις. Εάν θέλουμε όμως να μιλάμε για διαλειτουργικότητα, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για διαλειτουργικότητα τεχνικών συστημάτων και όχι νομικών συστημάτων. Γιατί η επαλήθευση ταυτότητας, ε, η επαλήθευση ταυτότητας έχει μέσα απολύτως τεχνικά. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Εκτελεστικής Επιτροπής επ' αυτού. Έχει αλλάξει λίγο οπτική γωνία από την ταυτοποίηση που είναι φιλοσοφικός όρος μάλλον αμφιλεγόμενος, δηλαδή ποια είναι η ταυτότητά μου, ποιος είμαι. Ε, αν έχει περάσει λοιπόν στην επαλήθευση ταυτότητας ε, και πώς σκέφτεται να δημιουργήσει αυτήν την ε, διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών που βεβαίως είναι κάτι το οποίο προσδοκούν όλοι οι πολίτες. Επίσης είναι σημαντικό και νομίζω ότι οι συνάδελφοι συμφωνούν μαζί μου. Είναι σημαντικό λέω να μην επιτρέψουμε ε, να ε, υπάρξει μια περιδίνηση προς τα κάτω ε, σε σχέση με τα ή e στάνταρ τα οποία έχει, έχουν ήδη κάποιες χώρες γιατί υπάρχουν χώρες όπως τη Γερμανία ή στην Αυστρία που ε, θέλουν ε, διαχωρισμό, ενώ άλλοι όπως ε, η Σουηδία ή το Βέλγιο που τα βάζουν όλα στο ίδιο καλάθι. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι η διαλειτουργικότητα θα αφορά μονάχα τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την επαλήθευση ταυτότητας και ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα διαλύσουμε όλα τα θεσμικά εχέγγυα τα οποία υπάρχουν σε κάποιες χώρες. Επίσης, με εκπλήσει και κάτι άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ε, η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας σημαίνει ότι ε, παρέχεται κάποια υπηρεσία και επομένως θα πρέπει εγώ σαν πολίτης να έχω τη δυνατότητα επιλογής. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τεχνική εναρμόνιση ε, σε επίπεδο τέτοιο που ο πολίτης, εγώ δηλαδή, να μπορεί να επιλέξει το επίπεδο ε, αυτό το οποίο θα του δίνει όμως και την ηλεκτρονική εμπιστοσύνη ε, που θα του δίνει πρόσβαση στο, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά δεν θα ε, μειώνει το επίπεδο ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης που έχει. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο εθίγει είναι το εξής πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια και τις εφαρμογές της. Και εγώ θα προτιμούσα, σαν Επιτροπή, να μιλήσουμε για ασφάλεια μέσω της διαφάνειας, δηλαδή ε, να μπορεί να, να γίνονται ε, ανεξάρτητοι έλεγχοι, να δεχόμαστε τον έλεγχο και τρίτον και όσον αφορά ε, και την ε, οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή του 1999 εκεί υπήρχε μια ε, ε, σοβαρή πολιτική ασφάλεια, η οποία όμως δεν έδωσε καμία όθηση στην οικονομία όπως ήταν η αρχική πρόθεση και επομένως εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των υπολείπων ε, πώς βλέπουν αυτήν την ιδέα της ασφάλειας ε, μέσω της διαφάνειας και πώς είναι δυνατόν να βάλουμε περισσότερα τέτοια στοιχεία σε αυτήν την οδηγία έτσι ώστε ε, και η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη να είναι μετρήσιμες, να μπορούν λογιστικά να ελεγχθούν και βεβαίως να οδηγήσουν σε διαλειτουργικότητα. Περιμένω κυρίως τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού και ευχαριστώ πάρα πολύ ε, όλους για τη συνεργασία και το χρόνο που αφιέρωσαν στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλον ε, ε, σκιώδη. Πρώτος εγγεγραμμένος βουλευτής, ο συνάδελφος Οντή. Παρακαλώ κύριε Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους ε, σκιώδεις εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων ε, για αυτήν την πάρα πολύ σοβαρή ε, εργασία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο άρθρο 10 δεχόμαστε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνη που προέρχονται από τρίτε χώρε μπορούν ε, να ασκήσουν την παροχή υπηρεσιών στην ενωσιακή επικράτεια. Ε, φαντάζομαι ότι το αντίστοιχο μπορεί να γίνει ε, και με τρίτες χώρες οι οποίες όμως θα πρέπει να δεχτούν στην επικράτειά τους τους δικού μας παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η βασική έννοια της αρχής της αμοιβαιότητας άρθρο 19. Πρότεινα στον κατάλογο των προϋποθέσεων για την άσκηση ε, παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης ε, να ε, τους υποχρεώσουμε να αρνηθούν ταυτοποίηση, μάλλον πιστοποίηση παροχής ε, για ε, υπηρεσίες τις οποίες υποπτευόμαστε παράνομες. Με τον τρόπο αυτό να αποφευχθούν ε, οποιοσδήποτε τρομοκρατικές ενέργειες, διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κτλ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον ε, να τους υποχρεώσουμε να, δεχτούν ότι εφόσον έχουν έστω και κάποιες υπόνοιες ότι η δραστηριότητα είναι παράνομη να αρνηθούν την πιστοποίηση. Όσον αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή, εγώ προτείνω να μην είναι ακριβώς ισότιμη με την χειρόγραφη υπογραφή, αλλά ε, να θεωρηθεί ως τεκμήριο ε, ισοτιμίας. Σε πολλά άλλα σημεία θα υπάρξει και τεκμήριο ισοτιμίας. Ε, νομίζω όμως ότι ο κίνδυνος απάτης είναι μάλλον μεγαλύτερος κατά την άποψή μου στα πλαίσια αυτής της ηλεκτρονικής υπογραφής παρά της χειρόγραφης υπογραφής. Και ε, εάν το θέμα φτάσει ενώπιον της δικαιοσύνης, ε, τότε την κυριαρχία κατά κάποιο τρόπο επί της ηλεκτρονικής θα έχει η χειρόγραφη υπογραφή. Να μην δώσουμε πλήρη ισοτιμία δηλαδή, τουλάχιστον για 5-6 χρόνια για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Τελευταία παρατήρηση και ευχαριστώ την συγγήτρια που το ανέφερε επί των ε, κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων και αυτό είναι μια γενικότερη σκέψη ε, κυρία Πρόεδρε ή με τρομοκρατεί ο τρομερός αριθμός κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων ε, που ε, ε, καλούμαστε να δεχτούμε στα πλαίσια αυτής της νομοθεσίας και των νομοθεσιών γενικώ που καλούμαστε να, να δεχτούμε. Όλη η νομοθεσία η οποία συνδέεται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με πάρα πολλές κατεξουσιοδότηση πράξεις, έστω και αν αυτές είναι ε, ε, υποχρεωτικές, γιατί καταλαβαίνουμε την ε, σημασία τους στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, αλλά πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο η λειτουργικότητά τους δεν είναι απολύτως συνδεδεμένη με την γενικότερη εργασία που κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Πρόεδρε, στη διάσκεψη των Προέδρων, να ζητήσετε αξιολόγηση των διοικητικών μέσων που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να ελέγξουμε πολιτικά τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, που δεχόμαστε, οι οποίες μπορεί να είναι απολύτως αιτιολογημένες, αλλά δεν μπορούμε να τις δεχτούμε εάν ε, δεν μπορούμε να ασκήσουμε και τον πολιτικό έλεγχο αυτών των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε, αγαπητέ συνάδελφε, θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό, ε, το οποίο μου φαίνεται απόλυτα, σωστό, στη διάσκεψη των Προέδρων. Ε, θα ζητήσουμε λοιπόν από την διάσκεψη των Προέδρων αυτή την αξιολόγηση των κατεξουσιοδότηση πράξεων που ζητάει ο συνάδελφος Όντι και που αφορά ε, και την παρούσα περίπτωση αλλά και άλλες. Τώρα, εάν δεν έχουμε άλλους συναδέλφους, ε, να δώσουμε το λόγο στον Ανδρέα Σερβίδα, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι περιμένουν με αγωνία να ακούσουν την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω ότι θα απαντήσει και στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και όλα τα εξάτιμα μέλη αυτής της Επιτροπής για τη συμβολή τους στην επεξεργασία και τη συζήτηση της πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Το σημείο εστίασης της εισηγήτριας για το τι ακριβώς θα επιτευχθεί, ποιος είναι ο μακροχρόνιος, ε, μακροπρόθεσμος στόχος της πρότασης, είναι ακριβώς αυτό που κινεί και εμάς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την επεξεργασία ε, ενδεχόμενων βελτιώσεων για την πρόταση. Ως ε, γενικές παρατηρήσεις, πριν περάσω στα ερωτήματα των μελών για τις τροπολογίες, πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τους ε, στόχους, την πρόθεση ε, των τροπολογιών. Βεβαίως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το γενικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα παραμείνει ε, στον ε, γενικό στόχο της ε, προαγωγής της εμπιστοσύνης και θα επιτρέψει σε όλους τους εταίρους να δράσουν με το ίδιο πνεύμα. Διασφάλιση ύψος του επίπεδου ασφάλειας, διαφάνειας στις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό. Βεβαίως και αναλογικότητα είναι σημαντική, ιδίω ε, σε σχέση με τα όσα προτείνονται ως ένα δεχόμενο καθεστώς για τους ε, παρόχους υπηρεσιών που είναι κατάλληλοι. Είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Και θέλουμε και εμείς να εργαστούμε μαζί σας για να μεριμνήσουμε ότι θα τηρηθεί αυτή η αρχή προ όφελο όλων των μερών και των παρόχων υπηρεσιών και των, ε, πελατών, των, συγγνώμη, των πολιτών. Τώρα, α περάσω στα ερωτήματα των ε, μελών. Πρώτον, πράγματι για την ε, επαλήθευση έναντι της ταυτοποίηση, Να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός δεν έχει την πρόθεση να εναρμονίσει τις τις διατάξεις που αφορούν ε, την ε, ταυτότητα και την ε, διαδικασία επαλήθευσης. Έχει ως στόχο να θεσπίσει ένα ελάχιστο νομικό καθεστώς που θα δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ηλεκτρονικών μέσων ταυτοποίησης, κάτι το οποίο παρέχεται ήδη στα κρατημέλη και το αναγνωρίζουν ήδη τα κράτη-μέλη. Και, είναι... και μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ε, μέσω αυτών των ε, εργαλείων. Όταν αυτό θα συμβεί, τότε τα κράτη-μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν ένα ή περισσότερα τέτοια προγράμματα που αναγνωρίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους για να δίνεται δυνατότητα πρόσβαση ε, στις δημόσιες υπηρεσίες εκτός της επικράτειας όπου παρέχονται αυτά τα μέσα. Ιδίω, γι' αυτό μας αφορά σε αυτόν τον κανονισμό, οι υπηρεσίες που, ε, στις, για τις οποίες απαιτείται η χρήση των ε, μέσων ε, ε, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Γι' αυτό και παρέχεται αυτό το νομικό πλαίσιο για να ενισχυθεί η τεχνική διαλειτουργικότητα με μια σχετική πλατφόρμα, κάτι το οποίο αναφέρθηκε από τον κύριο Κρούσμαν. Τώρα, για τις, δραστηριο... τις πιλωτικές δραστηριότητε που έχει χρηματοδοτήσει η Επιτροπή του 2008, ιδίως το πρόγραμμα STORK, Εδώ πράγματι μπορώ να σας πω ότι στόχος μας δεν είναι η αναμόνηση. Και η αναγνώριση, τα μέσα ε, ηλεκτρονικής αναγνώρισης συνδέονται ιδιαίτερα με τα ε, μέσα επαλήθευσης είναι το σημείο εστίασης για μας. Βεβαίως, οτιδήποτε κινείται προς αυτή την κατεύθυνση θα μας βρει σύμφωνος ο πλευράς Επιτροπής. Τώρα, ίσως μπορούν να υπάρξουν στοιχεία ε, καταχώρησης της ταυτότητας ε, που υπόκειται αποτελούν αρμοδιότητα του κράτους μέλους και δεν μπορούν να τύχουν εναρμόνισης από εμάς. Και όπως αναφέρθηκε, πράγματι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την πλήρη αρμοδιότητα για αυτή τη δραστηριότητα. Δεύτερον, για την επιλογή που έχει ο πολίτης. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την χρήση των ε, μέσων ηλεκτρονικής ε, ταυτοποίησης για την ε, πρόσβαση σε υπηρεσίες, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αυτή η ελευθερία επιλογής. Ακόμα και στον κανονισμό δεν αποκλείεται αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι η αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ε, θα πρέπει να δούμε τι επίπεδο και τι είδους μέσα θα έχουμε. Όλα αυτά αποτελούν πλήρη αρμοδιότητα ε, του, του, του πολίτη που θέλει να, να πάρει αυτή την ε, ταυτοποίηση. Πλέον υπάρχει υποχρέωση λοιπόν, πρόκειται για δημόσιες ε, αρχές ή για παρόχους δημοσίων υπηρεσιών που σε εθνικό επίπεδο έχουν αποφασίσει τι είδους ε, τέτοιου μέσου θα χρησιμοποιήσουν και τι επίπεδο ασφαλείας θα έχουν σε ό,τι φορά τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο κανονισμός λοιπόν δεν ε, αποκλεί ε, την, αυτή την, το ενδεχόμενο επιλογής, όμως υπάρχει και το ζήτημα τη ευθύνη των δημοσίων αρχών. Εκείνε πρέπει να επιλέξουν. Και είναι και αρμοδιότητα των κρατών μελών να εγκαθιδρύσουν κατάλληλα ε, προγράμματα για να δώσουν δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο σύστημα πιστοποίησης λοιπόν. Τέλος, για την ασφάλεια μέσω της διαφάνειας, να είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η αρχή και συμφωνούμε απολύτως ως Επιτροπή. Γι' αυτό, ιδίως για τους εγκεκριμένου ε, παρόχους ε, παλήθευσης, θα υπάρξει υποχρέωση για τους παρόχους πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους, αλλά και κατά τη διάρκεια πρέπει να έχουν και μια, ε, να υποβάλουν εκθέσεις για την ε, συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και θα πρέπει να διασφαλίζουν ασφάλεια, αξιοπιστία και συνέχεια ε, της ε, δράσης τους. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Μαρίτα Ουλσκοκ θα, ολοκλη... θα είναι η τελευταία να ολοκληρώσει τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε από τους προλαλήσαντες, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το σημαντικό αυτό οικοδόμημα και υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξει μια εναρμόνιση προς τα κάτω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα, κάτι το οποίο είναι απευκταίο. Η υποδομή που θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύπτει τα πάντα από την ελευθερία έκφρασης μέχρι την οικονομική ανάπτυξη και μια ανθούσα αγορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών Και θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η Κομισιόν. Λέγουσα ότι δεν πρόκειται μονάχα για μια εναρμόνιση, πρόκειται για τη δημιουργία διαλειτουργικών δομών. Τα συστήματα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν να κατανοούνται αμοιβαίω και να αναφέρονται το ένα στο άλλο. Αυτή είναι η βασική ιδέα που διατρέχει αυτό το νομοθέτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταυτίζονται στη δομή του Η πύλα έκανε μερικά εύστοχα στο σχόλια και συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπε. σε σχέση με το ρόλο των εποπτικών αρχών. Εκεί πρέπει να γίνουν σημαντικές πρόοδοι. Χρειαζόμαστε επίσης να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε σχέση με την εξέβρεση λύσεων για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό της ε, αδειοδότησης των υπηρεσιών εμπιστοσύνη και της έγκρισης των. Θα πρέπει να κρατήσουμε και σε ένα λογικό επίπεδο την γραφειοκρατία και τη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά χρειάζεται να εξασφαλίσουμε και η ασφάλεια μέσω των κανόνων. Τα σχόλια του κυρίου Κρότσμαν για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία επαλήτευση ταυτότητας, ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μας. Και χρειάζεται όμως παράλληλα να εξασφαλίσετε και το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό σημαίνει καλύτερο συντονισμό και με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για να καταλήξουμε σε ένα πιο πρόσφορο σύστημα. Για αυτά που είπε η Αμέλεια Άντερστότερ, δεν μπορούμε να έχουμε μια εναρμόνιση προς τα κάτω. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν αυτή η διαδικασία εναρμόνιση στο χαμηλό το κοινό παρονομαστεί. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των παρόχων από τρίτες χώρες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Βλέπω ότι πολλά από τα ερωτήματα αναφέρονται στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης όπου υπάρχει μεγαλύτερα βεβαιότητα για, το, για τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε, ενώ τα θέματα της ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας είναι εκεί που είναι σχετικά ίσονες οι διαφορές απόψεων και νομίζω ότι εκεί έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μεγάλη πρόοδο. Δεν θέλω τώρα να σας καταπονήσω με τεχνικές λεπτομέρειες, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι ο συντονισμός των προσπαθειών μας με την ΙΜΚΟ θα γίνει πιο έντονος από τη στιγμή που θα έχουν προχωρήσει και αυτοί στην επεξεργασία τους. Δεν μπορούμε να περάσουμε σε μια συζήτηση σε βάθος με την ΙΜΚΟ προς το παρόν, διότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε μαζί τους. Ευχαριστώ. Άψογα ολοκληρώθηκε η εξέλιξη του σημείου αυτού. Νομίζω ότι ε, ε, η συζήτηση έγινε με εξαιρετικό τρόπο, ταυτοποιήθηκαν τα, τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτού του ιδιαίτερος σημαντικού κανονισμού. 18 ε, Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην ομάδα μας, ενώ η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για το Δεκέμβριο του 2013. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό, προχωράμε με παρόμοιο θέμα. Ε, το η πρωινή μας συνεδρίαση ασχολείται πολύ με αυτά τα θέματα. Έχουμε το σημείο 5, έκθεση εφαρμογής σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια Κατρίν Τροτμάν, λέγοντάς σας εξ αρχής ότι θα έχουμε κάποιες ειδικέ παρεμβάσεις της Κομισιόν και κάποιων εκπροσώπων ρυθμιστικών αρχών ε, πριν πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Το λόγο έχει λοιπόν η Κατρίν Τροτμάν να μας κάνει την πρώτη εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώντας αυτήν την παρουσίαση της έκθεσης που πρέπει σήμερα μάλιστα να καταθέσω στην ε, προσμετάφραση, ε, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι θα ήθελα ιδιαίτερω να ευχαριστήσω τον κύριο Βιολάν, ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ε, ήρθε εδώ ήρθε εδώ για να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία απευθύναμε στην Κομισιόν. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Καράτσογλου και τον κύριο Ντετομάζο που εκπροσωπούν εδώ το Μπέρεκ και που επίσης έχουν κάνει εξαιρετική εργασία και για μένα ε, και για τους σκιώδεις εισηγητές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεσή μου δεν έχει ακόμα ε, ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα συζήτηση για το ακριβές περιεχόμενο, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια γενική συζήτηση ε, επί του γενικού περιεχομένου ε, και με μεγάλη προσοχή λοιπόν θα ακούσω τις απόψεις, ανησυχίες, προβληματισμούς, συστάσεις και συμβουλές των συναδέλφων και οδών εισηγητών. Υπενθυμίζω το διακύβευμα της εκθέσεως. Οι δέσμοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007 ε, έγιναν μακρύς διαπραγματεύσεις μέχρι το 9 έτσι ώστε να υπάρξει ταυτο, ε, συγγνώμη, ε, υλοποίηση στα κράτη-μέλη ε, και ενώ τον Μάιο του 11 προεβλέπεται η, η αρχική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει μερική ή εξολοκλήρωνα θεώρηση αναθεώρηση της δέσμης και το ερώτημα το οποίο θέτω εγώ εδώ είναι ότι ε, υπήρξαν πρόοδοι και ποιες είναι αυτοί και ε, υπάρχουν ελλείψεις ε, και επίσης να ταυτοποιήσουμε τις ελλείψεις. Ε, μαζί με τους δύο συναδέλφους που είμαστε οι τρεις σωματοφύλακες κατά κάποιο τρόπο των ε, τηλεπικοινωνιών, συγγνώμη, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ε, ε, ε, ε, είχαμε την άποψη ότι πρέπει η νομοθεσία να είναι τέτοια που να επιτρέπει την προβλεψιμότητα και την αποτελεσματικότητα αλλά να δίνει και την δυνατότητα αύξησης της συνρύθμισης και ταυτοχρόνως να μπορεί να μειώσει το διοικητικό βάρος το οποίο διαπιστώνουμε αναλύοντας τις αγορές και αυτή η, ε, αυτή η κίνηση χρειάζεται έτσι ώστε να απελευθερωθούν και να λειτουργήσουν καλύτερα οι αγορές. Αυτή την ισορροπία προσπαθήσαμε να βρούμε ε, ανάμεσα στον Μπέρεκ, σε εμά τους ίδιους, στον Μπέρεκ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Να κάνουμε λοιπόν μία αξιολόγηση, μία εκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη πώς έχουν τα διάφορα στοιχεία τώρα, να δούμε ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως είναι οι επενδύσεις, όπως είναι η ενίσχυση της νομικής ασφαλείας, πράγματα δηλαδή απολύτως απαραίτητα για την δημιουργία εμπιστοσύνης και επομένως ανάπτυξης ολόκληρου του κλάδου και ε, ακριβώς αυτό διαπιστώνουμε συζητώντας και με τις εμπλεκόμενες ε, εταιρείε. Επομένως δεν μιλάμε εδώ για ε, ένα θέμα το οποίο είναι στενά οικονομικό και αφορά στενά την οικονομική ρύθμιση, αλλά μιλάμε γενικότερα για την συνεισφορά που έχει, για τη συμβολή που έχει αυτός ο κλάδος στην γενικότερη αγορά. Και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και άλλωστε το είδαμε συζητώντας για την προηγούμενη έκθεση της συναδέλφου Ουλφοκ, ότι τα, θέματα της εμπιστοσύνης και της ε, νομικής ασφαλείας είναι ουσιώδου σημασίας εάν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά που όμως θα κινείται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όσον αφορά τα ρυθμιστικά μέτρα και όσον αφορά την τεχνολογία και όσον αφορά τις νομικές διαδικασίες. Έχουμε κάποιες θέσεις λοιπόν. Ε, είχαμε συζήτηση κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως προτείνει ας πούμε ε, η Κομισιόν ε, η δυνατότητα των επιχειρήσεων ε, να λειτουργήσουν ε, καλύτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής Επικράτειας, δηλαδή αυτό το θέμα της ταυτότητας. Επίσης το ζήτημα του φάσματος, αυτό είναι λιγότερο αμφίσιμο όσον αφορά το, τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, αλλά είναι πιο πολεμικό κατά κάποιο τρόπο εάν, σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Όπως έχουμε πει και συνάδελφοι το είπαν, θέλουμε να ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής σχετικά με τα θέματα τα οποία θέλει να τροποποιήσει και να προωθήσει. Πιστεύω ότι ιδίω μετά το RSPP η ε, Κομισιόν ε, λίγο έχει κάνει πίσω ας πούμε όσον αφορά το θέμα του φάσματος. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να πάρει θέση και νομίζω ότι σε σχέση με το φάσμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, τελικά απέπεμψε την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει το πάνω χέρι κατά κάποιο τρόπο στις ε, ε, διαπραγματεύσεις και επομένως μπορεί να προωθήσει διευρωπαϊκές υπηρεσίες. Επ' αυτού θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής. Ουδετερότητα του δικτύου και καθολική υπηρεσία και αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Συζητώντα την αναθεώρηση τη δέσμης, τα συζητήσαμε όλα αυτά. Η Κομισιόν μας είπε αφήστε τα τώρα, θα τα πιάσουμε αργότερα. Εντάξει, αλλά τώρα προκύπτει ξανά το ερώτημα. Ε, γιατί φοβούμε ότι εάν δεν υπάρξει πραγματική διαλειτουργικότητα θα έχουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες θα αφορούν ή θα είναι συνδεμένες με τεχνολογίες του παρελθόντος και άλλες οι οποίες θα συνδέονται ε, με ισχύουσες τεχνολογίες υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές. Το θέμα είναι σημαντικό κατά την άποψή μου και επομένως και από τον Μπέρεκ και από την Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογήσουν ε, την ε, ανάλυση του ορισμού των αγορών, ε, τις συμμετρικές και μη συμμετρικές δέσμες, το πλαίσιο δηλαδή γενικότερα ε, όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 και 7α, τα οποία πολύ συζητήθηκαν ε, και ορισμένοι ε, θεώρησαν ότι θα αποτύχουν οι διαπραγματεύσει από αυτόν, αλλά δεν έγινε όμως. Και νομίζω ότι όλα αυτά φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε λέγοντας, εκφράζοντας μάλλον για μία ακόμα φορά την ευγνωμοσύνη ε, προς τους ε, συναδέλφους. Ε, δυστυχώς δεν ήμουν στην τελευταία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν εξαιρετικά περίπλοκο και είχα και εγώ κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες δεν μου επέτρεψαν να είμαι παρούσα, αλλά οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα πιο έντονα όσον αφορά τις τροπολογίες και φυσικά θα λάβω υπόψη μου τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε πολύ για το εισαγωγικό σας σημείωμα. Τον ε, λόγο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν είναι ο κύριος Γιώλα εκπρόσωπο σήμερα, αλλά ο κύριος Άντωνη Βελάνα. Θα του δώσω αμέσως τον λόγο, παρακαλώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Συγήτρια και τα εξαρτημα μέλη του Κοινοβουλίου. Πράγματι, ο συνάδελφο ζητά συγγνώμη που δεν ε, μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Ή όπω είπε και η συγγήτρια όμω, ένταξε την ευκαιρία, την ευκαιρία για να ε, κοινοποιήσει κάποιε από τι απόψει του. Η συγγήτρια έχει θίξει σημαντικό αριθμό ζητημάτων. Χαίρομαι που και ο συνάδελφο εκ δεξιών μου είναι εδώ που είναι αρμόδιος για κάποια από αυτά τα ζητήματα και θα μπορέσει να σας απαντήσει στη συνέχεια. Το πιο θεμελιώδες ε, ζήτημα, πριν ε, διατρέξω κάποια από τα πιο συγκεκριμένα θέματα που ανέφερε η συγκήτρια, είναι το πώς να κάνουμε συμπεράσματα από την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι παρότι συμμεριζόμαστε την άποψη ε, ότι είναι λυπηρό που καθυστερεί τόσο πολύ η μεταφορά στα κράτη-μέλη της νομοθεσίας, νομίζω ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά όλα τα κράτη-μέλη τα έχουν, έχουν μεταφέρει στη την νομοθεσία, παρότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια θέση να Συμπεράνουμε λοιπόν ε, σε ένα επίπεδο για την λειτουργία του πλαισίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αρχίσουμε ήδη να συζητήσουμε σε βάθος τη γενική επισκόπηση του πλαισίου οδηγιών όπως ε, υιοθετήθηκε το 2009, εν μέρη εξαιτίας της ε, καθυστέρησης στην μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Όμως μπορούμε να συναγάγουμε κάποια ξεκάθαρα συμπεράσματα για ζητήματα που πράγματι πρέπει να αλλάξουν και τα οποία δεν ε, μπορούν να περιμένουν. Όπως έχει ήδη αναφέρει και η Αντιπρόεδρος Εκρούς... η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια κέρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής. Ήδη ανέφερε κάποια η εισηγήτρια στις παρατηρήσεις της, ιδίως το θέμα της εστίασης σε ένα μέσο διαβατηρίου για τη διευκόλυνση των διασυντηριακών δραστηριοτήτων των ε, τηλεπικοινωνιών. Και το ζήτημα του φάσματος έχει ε, αναζητηθεί. Λοιπόν, για την ιδέα του διαβατηρίου. Είναι ο ακρογωνιαίος λήθος ε, ε, στην, στο σκεπτικό του πακέτου της ενιαίας αγοράς. Ουσιαστικά η αδειοδότηση πρέπει να είναι μοναδική, ακόμα και για παρόχους που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες. Αυτό ε, ε, δημιουργεί αρκετή ε, ασφάλεια δικαίου έτσι κι όμως το αναφέρω ως ακραγωνιό λίθο γιατί με αυτή την αφετηρία Με αυτή την αφετηρία λοιπόν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και άλλα μέσα για να διασφαλίσουμε την πραγματική εναρμόνιση. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς κανονιστικούς τομείς σε ό,τι αφορά την ανάλυση της αγοράς έως και την προστασία των ε, τελικών καταναλωτών, ε, τελικών χρηστών και πολιτών σε ό,τι αφορά το, τη δέσμη ε, του 2009. Όμως Μπορεί να υπάρξει και δυνατή διαφοροποίηση στη βάση και έτσι είναι και παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η δραστηριοποίηση σε πολλές χώρες. Το σημείο εστίαση λοιπόν τη Επιτροπής με αυτή την ιδέα του διαπατηρίου είναι να εντοπίσουμε του τομεί όπου η ασφάλεια δικαίου των ε, ε, παρόχων μπορεί να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό με πιο εναρμονισμένους όρους χωρίς αυτό να έρχεται σε βάρος ε, των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Και η ίδια η απόκληση, αυτή η διαφοροποίηση ε, δημιουργεί ζημίες για όλους. Όμως η Επιτροπή σε οποιοδήποτε εγχείρημα αναρμόνισης θα πρέπει να έχει κατά νου την ανάγκη επαρκούς κοινού επίπεδου προστασίας που θα λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες των κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης εν συντομία να σχολιάσω το θέμα του φάσματος. Πρέπει εδώ να αποδώσουμε τα έψημα στο Κοινοβούλιο, στο πακέτο του 2009, υπήρξε το λεγόμενο launchpad που έδωσε κάποια ωφέλη σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας ε, της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρυζωνικό δίκτυο και προστασία άλλων ε, σημαντικών πολιτικών στόχων. Όμως θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι το RSPP μας έφτασε μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Ιδίως οι διατάξεις του που αφορούσαν την ευθυγράμμιση των όρων αδειοδότησης στα κράτη-μέλη. Ήταν ελάχιστες αυτές οι διατάξεις ό,τι αφορά την ε, ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εκεί θέλουμε να επικεντρωθούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγαλύτερο βαθμό στην πρόταση για την ενιαία αγορά. Η εισηγήτρια μίλησε για την δυνατότητα προώθησης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Και εμεί πιστεύουμε ότι ένα από τα κύρια σημεία σε ό,τι αφορά την κινητή τηλεφωνία, βεβαίω αφήνουμε κατά μέρο το ακαθόδε ζήτημα τη περιαγωγή, είναι η δυνατότητα των εμπορευομένων να έχουν πρόσβαση ε, ακριβώ αυτό το πιο σημαντικό ζήτημα, την παροχή ε, υπηρεσιών κινητή τηλεφωνία. Αν πάρουμε το ένα παράδειγμα μπορούσε να θεωρηθεί και πιο βολονταριστικό σε ό,τι αφορά τις ε, ε, δορυφορικές υπηρεσίες ε, κινητής τηλεφωνίας. Τα πιο σημαντικά επιτέγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε πολύ σημαντικό βαθμό είδαμε ότι επιτέθηκαν μέσω της υπονόμευσης των αποκλήσεων στα καθεστώτα αδειοδότησης στα κράτη-μέλη. Για, για τα ένδικα μέσα, η εισηγήτρια ανέφερε κάποια ζητήματα συμμετρικά έναντι ασημέτρων, ε, το, το δίλημα εξάντα Πράγματι, εμείς συμμεριζόμαστε τη φιλοδοξία της ε, εισηγήτριας να λειτουργήσει το πλαίσιο με έναν τρόπο που θα μας δίνει τελικά τη δυνατότητα άρσης ε, κανονιστικών περιορισμών. Είναι γνωστό ότι εμείς ε, θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα να προωθήσουμε λύσεις σε κανονιστικό επίπεδο που να δημιουργούν μεγαλύτερη σύγκληση, να διαμορφώνουν ε, σταθερό περιβάλλον επενδύσεων και ταυτόχρονα να έχουμε ε, ισχυρά ανταγωνιστικά εχέγγυα για να διατηρείται και η ευελιξία. Έτσι δεν άρουμε ουσιαστικά, δεν θα άρουμε το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά θα επαναπροσδιορίσουμε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Τώρα, για τη συνολική δομή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη σημασία της ε, του ασύμμετρου κανονιστικού πλαισίου βάσει της ε, ταυτοποίησης πραγματικών προβλημάτων της αγοράς με σημεία συμφόρησης και ούτω καθεξής. Στην αναθεώρηση των ε, αγορών, που είναι ένα εγχείρημα που έχουμε αναλάβει εκ αυτή είναι η βασική μας αρχή και δεν χρειάζεται να την αναθεωρήσουμε. Παράλληλα βεβαίως υπάρχει και νομοθετική πρωτοβουλία που έχουμε καταθέσει στο Κοινοβούλιο για την ε, διευκόλυνση των επενδυτικών δαπανών για τα βιζωνικά δίκτυα που ε, ενέχει περισσότερα συμμετρικά στοιχεία που ξεπερνούν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Χωρίς όμως να αλλάζει η γενική ισορροπία. Στην τελική ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την άποψη ότι το σήμα θα πρέπει να ενισχυθεί. Το, τα κανονιστικά πλαίσια τα εξάντα των εκ των, υστέρων, έχουν, των, εκ προτέρων έχουν έναν στόχο να ε, επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα και όχι το ευρύτερο πλαίσιο. Σε ό,τι φορά την, τις επαφές με τις εθνικές αρχές, για το άρθρο 7α με τη δημιουργία του Μπέρεκ και τη δική του συμβολή στις επιμέρους διαδικασίες, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά, αρκετά ικανοποιητικά, σε ό,τι αφορά τις επαφές μας με τον Μπέρεκ για τα ένδυγα μέσα. Στην πράξη λοιπόν είχαμε αγαστή συνεργασία και συνέκλυναν οι θέσεις μας στην μεγάλη πλειονότητα των ε, περιπτώσεων. Η ικανοποίηση δημιουργεί και το ότι στην μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων και πάλι, όπου έχουμε περάσει στην φάση 2 των ενδικών μέσων, έχει βρεθεί λύση βάσει της ευθυγράμμισης με την γνωμοδότηση Μπέρεκ, όπου ε, η Εθνική Αρχή είτε αποσύρει είτε τροποποιεί την πρότασή της. Στις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει σύσταση προς ε, την Εθνική Αρχή στο τέλος της διαδικασίας, τα αποτελέσματα είναι μεικτά, ανάμεικτα. Και αυτό δεν ε, μας εκπλήσει. Είναι μάλλον αφιλεγόμενος ε, ο τρόπος ε, που προτείνεται από το 7-7α. Ξέρω ότι δεν έχω καλύψει όλα τα σημεία. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Λοιπόν, όχι, νομίζω ότι Ήδη έχουμε μακρηγορήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω, όπως και η κυρία ε, Τροτμάν, τους δύο καλεσμένους μας, όχι γιατί εκπροσωπούν ε, αρχές, αλλά και γιατί έχουμε και ένα άνθρωπο που ήρθε την Ελλάδα, ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση σήμερα το πρωί και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Και εμείς. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο αμέσως στον κύριο Καρατζόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί την ETT, τα δηλαδή την Ρυθμιστική Αρχή της Ελλάδος, και μετά τον κύριο Ντε Τομάζο. Κύριος Καρατζόγλου, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας αναφέρω ότι και εγώ και ο κύριος Δετομάζο βρίσκονται εδώ εκπροσωπώντας τον ΜΠΕΡΕΚ, τον Φορέα των <clears throat> Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο Δόκτωρ Κανέλος, ο επικεφαλής της ΜΠΕΡΕΚ θα ήθελε πολύ να έρθει εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς κολλιόταν και δεν μπορούσε να αφήσει την Ελλάδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία αυτή την Ήτρε και την κυρία Τροτμάν ως εισηγήτρια για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου, για την ευκαιρία που μας έδωσε να παρουσιάσουμε τις κοινέ απόψεις των Ευρωπαίων Ρυθμιστών. Για το πλαίσιο υπήρξαν πρόοδοι μετά από την αναθεώρηση του 2009 και υπάρχουν και τομείς όπου μπορούν να επιτευχθούν περαιτέρω πρόοδοι. Οι απόψεις μας βασίζονται στην καθημερινή και απτή εμπλοκή μας στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Θέλω να τονίσω ότι η Μπέρεκ δεν έχει ακόμα επίσημο και εδρεωμένο, επίσημη συγγνώμη και εδρεωμένη θέση για αυτά τα αρκετά προωθημένα και παραστατικά θέματα. Επομένως θα χαιρετίζαμε ιδιαίτερα την ευκαιρία να συνεχίσουμε το διάλογο μας με τους Ευρωπαίους ρυθμιστές ως μια ευκαιρία να αναπτύξουμε περαιτέρω τον προβληματισμό μας είτε στα πλαίσια μιας γενικότερης αναθεώρησης είτε μιας πιο στοχευμένης παρέμβασης. Μετά από αυτήν την ε, σύντομη εισαγωγική παρέμβαση. Θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ντε Τομάσο για να προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένες απόψεις οι οποίες περιλαμβάνονται και στην έκθεσή μας προς την κυρία Τρότμαν που έχει η Επιτροπή σας στα χέρια της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωτού περάσω στο περιεχόμενο, θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω την κυρία Τρότμαν και την Επιτροπή Τρότμα, την Επιτροπή Ήτρα για την ευκαιρία αυτή να ανταλλάξουμε απόψεις με τις νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της σημερινής συζήτησης είναι να ανταλλάξουμε απόψεις για την καταλληλότητα του τωρινού πλαισίου για να αντιμετωπίσει τα τωρινά προβλήματα και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Η κοινή άποψη μέσα στην ΠΕΡΑΚ είναι γενικά θετική. Πιστεύουμε ότι το τωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές και μπορεί να παίξει και το ρόλο ενός μοχλού για σταθερότητα και συνεκτικότητα στο ρυθμιστικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μετά από το σαφές μήνυμα που μας έδωσε η κυρία Τρότμαν Θέλω να τονίσω ότι η τωρινή εργαλειοθήκη που έχουμε σε ρυθμιστικό επίπεδο είναι αποτελεσματική και κατανοητή από τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε σχέση με τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών. Επίσης, με τον τρόπο αυτό έχουμε δώσει τους εθνικούς ρυθμιστές εργαλεία σε πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, εργαλεία σε ό,τι αναφέρεται στη λειτουργική διαχώρηση και τη δυνατότητα να υπάρξουν ρυθμίσεις προς τον τομέα αυτό, την, την δυνατότητα να έχουν συμμετρική ρύθμιση όταν αυτό είναι απαραίτητο, εξασφάλιση της ουδετερότητας του διαδικτύου, ε, κατανομή του φάσματος και τα λοιπά μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα εργαλεία <clears throat> μας επιτρέπουν να προωθήσουμε λοιπόν το έργο των εθνικών ρυθμιστών. Γενικά λοιπόν είναι θετική η εκτίμησή μας. Θεωρούμε ότι η Μπερέκ έχει ήδη παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να εδραιώσει ένα Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Συμβούλιο και να προωθήσει μια κοινή ρυθμιστική ατζέντα σε όλη την Ευρώπη και θα είμαστε έτοιμοι και στο μέλλον να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο σε άλλα θέματα. Έχουμε ήδη με την καθημερινή μας εμπειρία εντοπίσει το μίσο που μπορούν να υπάρξουν πρόοδοι. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να μην προχωρήσουμε σε επαναστατικές αλλαγές, αλλά με σταθμιές μεταβολές να βελτιώσουμε το πλαίσιο που υπάρχει. Είμαστε έτοιμοι επίσης να παρουσιάσουμε την άποψη, τις απόψεις μας με πιο επίσημο τρόπο, εάν αυτό το θέλετε. Υπάρχουν πολλοί τομείς προβληματισμού για τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό σε ό,τι αφορά τους τερματικούς εξοπλισμούς και το ρόλο των παρόχων, το ρόλο των εθνικών διαδικασιών για κρατικές επιδοτήσεις, το μελλοντικό πλαίσιο της συμμετρικής ρύθμισης ή την ανάγκη να δούμε την ευρύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Will της Κομισιόν όταν αναφερόταν στην πρόταση της Κομισιόν για το κόστος της ε, δημιουργίας υποδομών. Όπως είπε και ο κύριος ε, Καρατζόπουλος, η Μπέρεκ δεν έχει μία άποψη ακόμα για τα θέματα αυτά, αλλά όταν έχουμε τέτοιες απόψεις θα σας τις διαβιβάσουμε με μεγάλη χαρά. Περνάω τώρα στα πια σημαντικά στοιχεία σκέψης. Για το άρθρο 7 εμείς συμμεριζόμαστε τις απόψεις της Κομισιόν και χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα που μπόρεσε να προκύψει από την συμμετοχή της Μπέρεκ στην ε, διαδικασία αυτή δημιουργίας κανόνων. Πιστεύουμε ότι η Μπέρεκ μπόρεσε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που της επέτρεπαν οι κανονισμοί να δώσει χρήσιμες και ανεξάρτητες ε, απόψεις για τα θέματα αυτά. Οι αποφάσεις που έχουν ε, ληφθεί μέχρι τώρα έχουν ε, σε όλους αυτούς που είχαν σκεπτικισμό για τη διαδικασία αυτή και είχαν ανησυχίες για τον έλεγχο ομοτήμων. Γενικά η Μπερέκα έχει υποστηρίξει τις απόψεις της Κομισιόν και στις λίγες περιπτώσεις που αυτό δεν έγινε. Αυτό ήταν φυσικό και δεν είχε παθολογικό χαρακτήρα γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Για το άρθρο 19, τη συνεργασία με την Κομισιόν και την εκπόνηση συστάσεων, εδώ υπάρχουν ίσως τομείς όχι βελτίωσης περισσότερο, αλλά διευκρίνησης, για να το πω καλύτερα. Μερικές φορές οι συστάσεις οι οποίες έχουν ε, εφαρμοστεί και συνεχίζεται ο έλεγχος για τη μη διάκριση και τη σωστή κοστολόγηση, υπάρχουν ορισμένα μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εργασιακές συνθήκες που δεν είναι πάντα εύκολο να ληφθούν υπόψη μέσα στη ρυθμιστική αυτή διαδικασία. Πιστεύουμε επίσης ότι η εφαρμογή αυτών των συστάσεων μπορεί να δώσει στην Κομισιόν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το άρθρο 7 και να λάβει περισσότερο υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες όταν ερμηνεύει αυτές τις συστάσεις. Για την ε, εκ των ε, ρύθμιση Επαναλαμβάνω αυτά που είπε η Κομισιόν, συμμεριζόμαστε απόλυτα την προσέγγιση αυτή. Ο κύκλος ρύθμισης είναι της τάξης των 25 ετών και βλέπουμε ότι υπάρχει μια βαθμία επίλυση των προβλημάτων και η Κομισιόν επεξεργάζεται τώρα ένα νέο κατάλογο θεμάτων που πρέπει να ρυθμιστούν. Και στο μέλλον μπορούμε να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και μας ενδιαφέρει όχι μόνο το θέμα της επέκτασης όλων αυτών των υπηρεσιών στις εποχές της υπαίθρου, αλλά θεωρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μια άντε αντιμετώπιση θα μπορούσε να είναι πιο αντιπροσωπευτική, πιο αποτελεσματική από τον έλεγχο μόναχα εξ το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως την ε, ύπαρξη πλήρους ανταγωνισμού. Επίσης προσπαθούμε μέσα στην ΠΕΡΕΚ να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά και χαιρόμαστε και για την ε, επισκόπηση και μεταρρύθμιση των ε, ρητρών οικουμενικής παροχής υπηρεσιών. Είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Κομισιόν και να συμμετάσχουμε περαιτέρω. Εν κατακλείδη είναι γεγονός ότι το τωρινό σύστημα συνρύθμισης μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών λειτουργεί πολύ καλά. Χρειάζονται βέβαια κάποιες βελτιώσεις στο επίσημο σύστημα επισκόπησης και αναθεώρησης προτού αυτό το σύστημα εφαρμοστεί πλήρως. Παραδείγματος χάρη, είναι χρήσιμο όταν υπάρχουν επανειλημμένες περιπτώσεις στοιχείων που προκύπτουν από τις εθνικές αναλύσεις εδώ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα και σε επίπεδο ουσίας νομίζω ότι είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία και στην πράξη το θέμα του ύψους, του, του άκτους μάλλον, του βάρους απόδειξης είναι κάτι που παραμένει πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ ψηλό αυτό το άκτος. Ένα τελικό μήνυμα από τη δική μας πλευρά μας ενδιαφέρει η νέα θεσμική δομή για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ανεξάρτητα και μέσα στην ΜΠΕΡΕΚ. Χαιρόμαστε πολύ για το τωρινό σύστημα που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Το πλαίσιο του 2009 μας εξασφαλίζει ένα σαφή ορισμό της ανεξαρτησίας και λειτουργικής και διοικητικής και έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την ανεξαρτησία των εθνικών αρχών από την πολιτική. Όταν φτάσουμε τώρα στην εφαρμογή σε εθνικό πλαίσιο υπάρχουν όπως ξέρετε ευκαιρίες και δυνατότητες για αναθεώρηση από τις εθνικές αρχές και εξαρτάται από την Κομισιόν να επισκοπεί και να επαληθεύει την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της ανεξαρτησίας. Για το μέλλον τώρα, νομίζουμε ότι το να υπάρξει μια πιο προσεκτική ματιά στην θεσμική αρχιτεκτονική των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για να καθοριστεί καλύτερα ο κέριος ρόλος τους και οι αρμοδιότητές τους. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ρυθμιστική συνεκτικότητα. Μας ενδιαφέρει επίσης να έχουν οι φορείς αυτή τη δυνατότητα για ένα πλήρη έλεγχο των πόρων τους. Μιλάμε για προπολογισμό, για ανθρώπινο δυναμικό και για την οργάνωσή τους. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να εξασφαλίσουμε ότι ο συντονιστικός ο ρόλος μας στην ΜΠΕΡΕΚ θα είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν μαζί σα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σα μεταφέρω και σα ευχαριστώ τα μάλλον. Χωρί μικρόφωνο η πρόεδρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρατζόγλου, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντετομάζο. Θα ξεκινήσουμε με του ε, ε, ε, ε από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε την εισηγήτρια ε, και... Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι η συγγετριά μας. Ε, ε, της έχω εμπιστοσύνη για την όλη διαδικασία και ευχαριστούμε πολύ και για τα όσα μας είπαν οι εμπειρογνώμονες. Άκουσα λοιπόν όλα αυτά και θυμάμαι ένα, μια παροιμία που λέγαμε παλιά ότι η εγχείρηση σε πέτυχε ενώ ο ασθενής απέθανε. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως λέει και η Επιτροπή, ε, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο, αλλά εγώ αμφιβάλλω κατά πόσον ουσιαστικά έχει μεταφερθεί η ε, νομοθεσία αυτή. Ε, κρίνω εκ των αποτελεσμάτων. Όταν, αποφασί, όταν πήραμε τις αποφάσεις για τις ε, τροποποιήσεις που θα έπρεπε να ε, λάβουν χώρα όσον αφορά τη δέσμη των επικοινωνιών, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. 50 εκατομμύρια κάτοικοι στην Νότια Κορέα έχουν ε, περισσότερες συνδρομές 4G από ό,τι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια και στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα πω ότι έχουν 20 φορές ε, ε, ψηλότερο επίπεδο ε, συνδέσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει το φάσμα τους είναι πολύ ευρύτερο. Τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα... Έχουν ακόμα συνδέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διαφορά των υπηρεσιών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Κομισιόν ε, λέει ότι έχει ε, μεταφερθεί στην εθνική, στην εθνική νομοθεσία η ενωσιακή νομοθεσία, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα μεγάλη κατάτμιση της αγοράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό στην ε, αναθεώρηση, γιατί η ίδια η δέσμη δεν ήταν αρκετή και αυτό είναι η μία σκέψη. Η άλλη σκέψη είναι ότι και ο τρόπος ε, υλοποίησης δεν είναι ικανοποιητικός κατά την άποψή μου. Βλέποντας πολλά στοιχεία, ε, ας πούμε η ε, απρόσκοπτη πρόσβαση σε τοπικά loops. Και εδώ έχουμε πρόβλημα. Και είναι σαφές ε, ότι δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα. Το unbundling ήταν μία από τις προϋποθέσεις και σαν αρχή αλλά και σε σχέση με τη διασύνδεση με, τις τοπικές, με, τους, ε, με τα τοπικά loops, τους βρόχους. Ε, θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση αν είχε χρησιμοποιηθεί πραγματικά όλο το οπλοστάσιο το οποίο ε, ε, υπήρχε βάση της νομοθεσίας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία έτσι ώστε να αλλάξει η πραγματικότητα επιτόπου. θα πρέπει να δούμε, να έχουμε τη γενικότερη εικόνα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως ε, συνδέεται και με την υλοποίηση του προγράμματος ε, φάσματος. Εδώ ξέρουμε ότι είναι λιπέστατη η υλοποίηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας πει εάν θα προχωρήσουν γιατί όλες ε, οι, όλα τα αιτήματα για ε, εξαιρέσεις ε, εξαιρούν θέσεις εργασίας, εξαιρούν την ανάπτυξη κυρίως. Μιλάμε για έναν τομέα ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη. Νομίζω και άλλωστε και η κυρία Τροντμάν το είπε και ο κύριος Γουλενάνης. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα με τις πανευρωπαϊκές αδειοδοτήσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα υπάρξει ενιαία, πραγματικά ενιαία αγορά εάν δεν δοθούν αυτές οι άδειες. Όλα τα άλλα θα συνεχίσουν τον κατακαιρματισμό της αγοράς που μπορεί να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος θα εξακολουθήσει πάντως να υπάρχει και θα σημαίνει ότι η αγορά είναι κατακαιρματισμένη. Και αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό για την Ευρώπη και για τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που της δίνει η ψηφιακή τεχνολογία και για να υλοποιήσουμε την εσωτερική αγορά και για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και σε ένα, άλλο, σε, σε ένα σωρό άλλα στοιχεία είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό αυτό που είπα προηγουμένως ε, και το θέμα της ηγεσία που πρέπει να κρατήσουμε όσον αφορά την τεχνολογία και τις επιστήμες όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Επίσης, ε, σημαντικό είναι να υπάρξει συνέχιση, follow-up και, αυτό θα, και θα επανέλθουμε σε αυτό και το είπα άλλωστε και στην εισηγήτρια. Δηλαδή, ότι τώρα πρέπει να δούμε εάν η στόχευση που είχαμε ε, με τον κανονισμό έχει υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Όπως είπα, η Κομισιόν λέει και ορθώς λέει ότι εφαρμόστηκε, μεταφέρθηκε στην Εθνική Νομοθεσία η δέσμη ε, για τις επικοινωνίες αλλά εγώ βλέπω ότι η πραγματικότητα δεν έχει καθόλου αλλάξει, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θέλαμε όταν ε, ε, υλοποιούσαμε την δέσμη Telecom. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να οθήσει την οικονομία της. Και επομένως, ένα είναι το ερώτημα. Πώς βλέπουμε τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που θέλαμε <coughs> να επιτύχουμε με τη δέσμη των ε, τηλεπικοινωνιών και τι, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα εκεί έξω. Η Ευρώπη δεν είναι ηγέτιδα δύναμη πλέον σε αυτό. Έχει μια κατακαιρματισμένη αγορά, ε, η οποία έχει μείνει πίσω, γιατί είναι πολλά μέρη της υφηλίου που προχωρούν με πιο γοργό βήμα. Και επομένως θα πρέπει να το ε, συζητήσουμε αυτό. Και επομένως στην αναθεώρηση θα πρέπει αφενός να διαπιστώσουμε με στοιχεία αυτό που λέω τώρα και αφετέρου να ε, ε, ενδυναμώσουμε την ανταγωνισμό για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο Φόκμαρ. Ε, ο Σένφος Σλότερ έχει το λόγο. Ή, ή συνάδελφος. Δεν ξέρω τι είδου σχόλια πρέπει να κάνω εδώ. Οπότε δεν θα σχολιάσω τίποτα. Ε, Ωραία, δεν έχουμε άλλους σκιώδεις, επομένως ε, τα μέλη της Επιτροπής να μιλήσουν. Ο συνάδελφος Κρότσμαν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και όπως είπε και ο συνάδελφος Φίγμαϊρ, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή άδεια για τους παρόχους των επικοινωνικών υπηρεσιών. Όμως το ερώτημα είναι, είναι έτοιμα τα κρατήματα για κάτι τέτοιο. θα, μπορούσαμε, θα μπορούσε αυτό ε, να οδηγήσει στην αποφυγή των χρεώσεων για περαγωγή, όμως παρόλα αυτά ε, τα κράτη-μέλη θα επιμείνουν οι άδειε να δίνονται στο δικό τους κράτος μέλος και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι βεβαίως πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Και εκ μέρους του κ. Βάλτιο να πω δύο πράγματα για την εφαρμογή του ε, πακέτου τηλεπικοινωνιών. Η συνάδελφος χαιρετίζει ε, την, ε, ε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και φαίνεται ότι αυτό το θέμα βρίσκεται επικεφαλής ε, στο θεματολόγιο της Επιτροπής. Χαιρετίζει και την ε, ανακοίνωση του προγράμματος για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς, της ενιαίας αγοράς Εν τω μεταξύ, έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε πώ έχει η κατάσταση σήμερα σε αφορά την εφαρμογή του τρίτου πακέτου των επικοινωνιών, την αποτελεσματικότητά του και να δούμε τι μπορούν να γίνει στο μέλλον. Καταλήγουμε όλοι στα ίδια συμπεράσματα. Ο τρόπο απελευθέρωση των αγορών έχει ωφέλη για του καταναλωτέ και αυξάνει και τον αριθμό των διαφορεμένων μερών στα 27 κράτη-μέλη, αλλά ενισχύει και τον κατακαιρματισμό ε, της ε, αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η φιλόσοφία είναι ότι η ε, παροχή περισσότερων αδειών και η αύξηση των ε, επιπέδων θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές. Επιπλέον, η εφαρμογή του πακέτου τηλεπικοινωνιών υπόκειται και στην ερμηνεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και έχει εφαρμοστεί με 20 διαφορετικούς τρόπους. Όσο εκ τούτου, το κόστος για τους παρόχους που δραστηριοποιούνται σε πολλά κατημέλη έχουν πολλαπλασιαστεί και δεν υπάρχει δυνατότητα για οικονομία κλίμακας. Υπάρχει λοιπόν ρυθμιστική αβεβαιότητα η οποία δεν ενθαρρύνει, ε, δεν οδηγεί σε περισσότερες επενδύσεις που είναι απαραίτητες και δεν καθιστούν τον τομέα της πληροφορικής έναν, ε, μια, ένα κριτήριο μοχλό για την ανάπτυξη. Πρέπει να διευκολύνουμε τους παρόχους στη δραστηριοποίησή τους σε διασυνορικό επίπεδο. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις να ε, μεγαλώσουν και να επανεπενδύσουν τμήμα των εσόδων τους. Αυτό θα μας οδηγήσει και στην ανάπτυξη ε, και στην καινοτομία ο τομέας πληροφορικής θα πρέπει να συνεχίσει να ε, κινεί ε, την οικονομία μας όπως έχει κάνει και την τελευταία δεκαετία. Η τεχνολογική καινοτομία και η τεχνολογία της ε, πληροφορικής θα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε και νέες προκλήσεις μπροστά μας, μπορούν να αποτελέσουν όμως ευκαιρίες θα μας ε, βοηθήσουν να αναθεωρήσουμε την διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής μας. Πρέπει να δούμε πώς, ε, κατά πόσο το κανονικό, κανονιστικό μας πλαίσιο μας επιτρέπει να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις. Ίσως να πρέπει να αλλάξουμε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Η ενοποίηση, όπως ε, δείχνει και το μοντέλο των ΙΠΑ, ε, βοηθά την ε, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, παρέχει κίνητρα για τους επενδυτές, διαμορφώνει ένα ειδικό οικοσύστημα επενδυτικό και διασφαλίζει ότι υπάρχει, θα υπάρξει μείωση κάποια στιγμή στις τιμές, όπως στο κόστος της Υπάρχουν προκλήσεις, όμως θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και έτσι μπορεί και η Ευρώπη να γίνει αποδοτική. Και αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό ε, σημάδι εν μέσω κρίσης. Αυτή ήταν η δήλωση της συναδέλφου την οποία ήθελα να σας μεταφέρω. Ευχαριστώ πολύ τον ε, συνάδελφο Κρότσμαν που πήρε το λόγο ε, εξ ονόματος συναδέλφου Βαλεάν. Συνάδελφοι, να, τώρα θέλετε το λόγο, πολύ ωραία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί φυσιολογικά οι φιλελεύθεροι λαμβάνουν το λόγο πριν από μένα. Γι' αυτό ένιωσα έκπληξη που μου δώσατε το λόγο. Δεν ήθελα να πάρω τη σειρά του κύριου Κρότσμαν. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποια σχόλια για την πανευρωπαϊκή διαδικασία αδειοδότησης. Υπάρχουν φορείς που εργάζονται και στην κεντροανατολική Ευρώπη, στην ε, Ολλανδία, σε άλλες χώρες. Υπάρχουν πολλές φορές μονοπόλια τοπικού χαρακτήρα. Οι κρατικές, ε, κρατικοί φορείς, οι τοπικά μονοπόλια, τα οποία όμως καλύπτουν ένα πολύ μικρό αριθμό πολιτών σε σχέση με το σύνολο των ε, πολιτών και καταναλωτών στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να σκεφτούμε για το θέμα των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια πρόκληση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο σαν μια αγορά για όλα αυτά τα προϊόντα, ενώ συγχρόνως διατηρούμε τις μικρότερες αγορές όπου μπορεί να υπάρξει ένα μικρό λειτουργικά μονοπόλιο το οποίο δεν επηρεάζει τη συνολική αγορά. Υπάρχουν εδώ ορισμένα σχέδια τα οποία προχωρούν στα κρατημέλη. Στην Βαρκελόνη, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν δίκτυα τα οποία λειτουργούν εκ των κάτω και λειτουργούν από τις τοπικές κοινότητες. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στη Βιέννη, στην Αθήνα, στο Βερολίνο. Χρησιμοποιούν τμήματα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για άλλες δραστηριότητες όπως είναι η κινητή τηλεφωνία ή ε, για επικοινωνίες σε επίπεδο τοπικό. Πέραν λοιπόν του τμήματος του φάσματος που έχει τύχει αδειοδότησης υπάρχουν πάντα δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί τμήμα αυτού του φάσματος για εθελοντικές δραστηριότητες που λειτουργούν με την θέληση της ίδιας τοπικής κοινότητας. Στο Άμστερνταμ παραδείγματος υπάρχουν τέτοιες εκπομπές που γίνονται με το τμήμα αυτού του φάσματος. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ληφθεί υπόψη ότι ένα τμήμα του ραδιοφάσματος μπορεί να χρησιμοποιείται για τέτοια τοπικά, για τέτοιες τοπικές πρωτοβουλίες και όχι να πηγαίνει στη γενική δυνατότητα κατανομής του φάσματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές φορές τίθενται και θέματα ασφάλειας και επομένως τα κράτη-μέλη δεν δέχονται να υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα δίκτυα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σύντομο σχόλιο προς τον κύριο Κρότσμαν. Ρώτησε, είναι έτοιμα τα κράτη μας μέλη για αυτό. Και το ίδιο ερώτημα μπορεί να τεθεί για οποιαδήποτε μεγάλη μεταρρυθμίση που έχουμε κάνει. Ήμασταν έτοιμοι για την ενιαία αγορά ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο πακέτο τηλεπικοινωνιών που τώρα το έχουμε συζητήσει. Αυτό το οποίο προέχει είναι να έχουμε μια σαφή εικόνα για όλα αυτά και να μπορούμε να συζητήσουμε για το αν αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση ή όχι ή να μείνουμε στα αυγά μας. Νομίζω ότι πάντα πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση εάν δεν παραμένουμε εκεί που είμαστε. Η ικανότητα λοιπόν να εξασφαλίσουμε την αλλαγή βρίσκεται στο να μπορούμε να συζητούμε για τα θέματα αυτά. Ορισμένε φορέ εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι όχι μόνο η πολιτική αλλά ακόμα και η τεχνική έχουν παραμείνει στο πλαίσιο της παλιάς τεχνολογίας. Και όταν μιλάμε για τα πανευρωπαϊκά πανευρωπαϊκή αδειοδότηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι παντού η ίδια συχνότητα. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό στις ΗΠΑ, αλλά όλα αυτά συνδέονται με κάποια διαδικασία αδειοδότηση. Νομίζω λοιπόν ότι με ένα καλύτερο συντονισμό μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση των ε, συχνοτήτων. Μπορούμε να είμαστε πραγματιστές και οραματιστές συγχρόνως το σημείο εκκίνησή μα όμω θα πρέπει να είναι η πραγματικότητα που είναι ότι σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου προχωρεί αυτή η διαδικασία πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν πιο γρήγορα βήματα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο Άκμαρ. Πολύ σύντομα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει στα ερωτήματα των ε, σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ ε, και τους ε, αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλια τα οποία και τις ερωτήσεις που απέφθηνα στην Κομισιόν. Θα ξεκινήσω με το σημείο το οποίο αφορά τις αδειοδοτήσεις του φάσματος. Ο κύριος Σόκβαρτ στη δεύτερη παρέμβασή του αναφέρθηκε ε, στο γεγονός ότι ε, πανευρωπαϊκή προσέγγιση δεν σημαίνει ε, μια μεγάλη αλλαγή, ένα, ένα big bang. Το, νομίζω ότι ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, όπου θα παίζει μόνο ένας πρωταγωνιστής. Δεν νομίζω ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι είναι έτοιμοι ή έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Αυτό που είναι σημαντικό για να φτάσουμε βαθμιδών στο σωστό δρόμο είναι οι πάροχοι ε, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ε, την παρέμβασή τους, την παρουσία τους σε πολλές χώρες, ε, γνωρίζοντας χρονοδιαγράμματα, γνωρίζοντας ε, τον τρόπο και τη διάρκεια των αδειοδοτήσεων. Αυτή είναι η σκέψη της ε, Κομισιόν και με τον τρόπο αυτό η διαδικασία θα είναι πιο αποτελεσματική κατά την άποψή μας. Οδηγούμε τώρα σε μία σε ένα άλλο σχόλιο. Είναι όντως σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο, το business model δεν είναι ένα ε, και βεβαίως ότι το φάσμα ε, της κινητής τηλεφωνίας δεν είναι το μόνο. Πρέπει να υπάρχει ε, ευελιξία ε, έτσι ώστε να βοηθηθούν ε, και όλοι ε, αυτοί οι οποίοι με τους δικούς τους, δικούς τους routers μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ελεύθερο φάσμα. Αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε ότι θα πρέπει, συμφωνούμε δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελεύθερο διαθέσιμο φάσμα το οποίο θα διέπεται από κάποιο πλαίσιο. Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ και με κάποιες άλλες ε, ερωτήσεις όσον αφορά το φάσμα πάντα. Σχετικά με το RSPP, η Κομισιόν βεβαίως ε, είναι εξίσου απογοητευμένη με την έκβαση της ε, κατάστασης Ναι, οι διερμηνείς ε, όντως παραπονούνται γιατί πρέπει να βγάλετε τα ακουστικά σας, είναι πολύ κοντά και να φέρει το μικρόφωνο είναι δυνατόν πιο κοντά στο στόμα του ο για να τον ακούμε καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα ε, του ε, ε, ε, των ελεύθερων ε, την ζώνη των 800 αυτό είναι θέμα διοικητικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για να δει κατά πόσον υπάρχει νομική συμμόρφωση όσον αφορά τις εξαιρέσεις να πούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ε, όντως πρέπει να υπάρξουν εκτός των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, έλεγχοι που αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με τρίτες χώρες και όπου είναι θεμητές διαδικασίες, αλλά οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της Κομισιόν επιμένουν στην ελαχιστότητα ταυτοποίηση αυτών των εξαιρέσεων ε, υπό το φως των ε, περιορισμών που υπάρχουν στον κλάδο. Και ελπίζουμε ότι ε, θέλουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος των ετοιμάτων εξαίρεσης μέχρι το καλοκαίρι όσον αφορά τις fixed markets και όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση. Βεβαίως ε, υπάρχουν πολλές διαφορές ε, στα κράτη-μέλη. Θα περίμενε κανείς ε, ότι αυτό το μοντέλο να είναι λιγότερο παρόν σε χώρες με αναπτυγμένη την καλωδιακή όμως ε, ε, ε, δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από αυτό το στοιχείο η διακύμανση. Η Κομισιόν έχει κάνει πάρα πολύ προσπάθεια όσον αφορά τις μη διακριτικές προϋποθέσεις και όσον αφορά την σύγκληση των τιμολογίων. και επομένως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε μέσω αντικειμενικών στοιχείων αυτήν την ε, διακύμανση που υπάρχει ε, στις ε, χώρες, ούτε εξηγείται μονάχα με οικονομικούς όρους. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση και πιστεύουμε ότι οι πάροχοι στις ε, διάφορες χώρες έχουν συγκεκριμένες ε, ανάγκες, ε, έχουν επίσης άλλες τεχνικές επιλογές για την πρόσβαση όσον αφορά είτε το virtual unbundling ή οποιαδήποτε άλλη virtual πρόσβαση στο δίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που δώσατε. Ο κύριος Καρατζόγλου και ο κύριος Ντετομάζο, εκπρόσωποι του Μπέρεκ, θέλουν να κάνουν επιπλέον σχόλιο, λαμβάνοντας υπόψη την συζήτηση την οποία παρακολούθησαν. Κύριος Καρατζόγλου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα, ο Μπέρεκ έχει επίγνωση ε, της πρωτοβουλίας για την ενιαία αγορά. Είμαστε ανοιχτοί και διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο κ. Ντεντομάζο, ο Μπέρεκ έχει εργαστεί στο θέμα της ε, μείωση του διοικητικού άκθου για τους πανευρωπαϊκούς ε, παρόχους. Και σίγουρα πρέπει να σημειωθούν περαιτέρω βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα από τα κύρια ζητήματα αφορά ε, τον καταγραμματισμό της αγοράς. Δεν είμαστε απεσιόδοξοι σε αυτό το θέμα. Υπάρχει όλο και περισσότερη εναρμόνιση που συχνά ενισχύεται και από συστάσεις της Επιτροπής. Αυτό βεβαίως αφορά περισσότερο τις ε, πιο όριμες αγορές αλλά όταν περνάμε σε αγορές νέας γενιάς με διαφορετικές ε, συνθήκες, ε, διαφορετικές συνθήκες αγοράς στα επιμέρους κράτη-μέλη σίγουρα επηρεάζουν τις εξελίξεις. Η Ευρώπη είναι μια νέα αγορά, αλλά έχουμε την Αυστρία για παράδειγμα, με πολύ σημαντικό διατροπικό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ε, ε, κινητού ευρυζωνικού δικτύου και σταθερού ευρυζωνικού δικτύου που ε, επιβάλλει στην ρυθμιστική αρχή να, να, βάλει πολύ συγκεκριμένες, να καθορίσει συγκεκριμένε τιμέ, γιατί αλλιώ δεν θα υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα ανταγωνισμού. Ενώ στι κάτω χώρε έχουμε ανταγωνισμό, αλλά υπήρξαν ε, και κάποια ζητήματα. Έχουμε την Ελλάδα, όπου μπορεί να μην είναι βιώσιμο, ε, χρήση των ινών μέχρι του, ε, τα σπίτια για μεγάλα ε, κομμάτια της χώρας. Λιθουανία, όπου η έλλειψη της αποσύνδεσης στο χαλκό έχει οδηγήσει τη χώρα να περάσει σε ε, δίκτυα FTTH και μάλιστα είναι μία από τις ε, κύριες δυνάμεις σε αυτό το τομέα, Σουηδία, όπου μικρά τοπικά προγράμματα έχουν οδηγήσει στην ε, κατακόρνη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH και ούτω καθεξής. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς όμως ε, να λαμβάνουμε υπόψη και τις ε, διάφορες ε, συνθήκες. Αυτό θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε καλύτερα στην κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Δετομάσο δεν επιθυμεί να παρέμβει. Ωραία, θα δώσουμε ξανά το λόγο στην Κατρίνα Τροτμάνα, έτσι ώστε να κάνει μια σύνθεση και να εξάγει συμπεράσματα. Είπαμε ότι η Κατρίν Τροτμάν ε, ήταν η συγγήτρια και της δέσμης ε, των τηλεπικοινωνιών. Είναι μέγας εμπειρογνώμων. Λοιπόν, ε, στις 9 Ιουλίου θα ψηφιστεί το θέμα στην Ήτρε και θα, σήμερα θα κάνουμε απλώς ένα προσωρινό κλείσιμο της συζήτησης. Κατρίν Τροτμάν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την Κομισιόν και τους εκπροσώπους της ΜΠΕΡΕΚ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που χωρίς καμιά αμφιβολία έχει εμπλουτίσει τον προβληματισμό μας και θα εμπλουτίσει και την εκθεσή μου. Θέλω να απαντήσω εν συντομία σε ορισμένε από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει, χωρίς τώρα να καλύψω όλα τα στοιχεία, αλλά θα ήθελα να δω ορισμένες θεματικές ενότητες. Καταρχήν, αν η ρύθμιση μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αγορά και να εξασφαλίσουμε ότι καταργούνται οι φραγμοί μεταξύ των 27 κρατών μελών. Η απάντησή μου είναι όχι. Θα βοηθήσει η ρύθμιση, αλλά δεν είναι το μόνο μέσο. Είχαμε προβλήματα και με τις αρχές ανταγωνισμού, έχουμε προβλήματα και με τις αρχές αντιοδότησης για το φάσμα συγνωτήτων. Πολλά προβλήματα τα οποία θα μπορούσα να σας αναφέρω. Είναι απαραίτητο η συζήτηση να είναι επακριβής ε, απτή και λειτουργική. Όλοι αυτοί οι οποίοι περεμβαίνουν στα θέματα της αγοράς και ιδίως σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση και τη λειτουργία της ρύθμισης αλλά και για τις επενδύσεις μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε μια άποψη τα θέματα αυτά. Πρέπει επίσης να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν πιστεύω ότι από μεθοδολογική έποψη για τους φορείς που λειτουργούν αυτές τις υπηρεσίες είναι θετικό να έχουμε ε, συνεχείς μεταρρυθμίσεις εμβαλωματικές χωρίς να εξασφαλίσετε η γενική συνεκτικότητα των ενεργειών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Μας ε, συγκρίνεται με τις Κορέες και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Μα είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κορέα υπάρχει μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο και ακολουθούν οι επενδύσεις και στην ε, ΗΠΑ Πολιτείε υπάρχει μια συνεργασία σε εδαφικό επίπεδο. Υπάρχει ένα είδος καρτέλ, όπως τα λέγαμε παλιότερα. Το ευρωπαϊκό σύστημα λοιπόν δεν είναι το ίδιο. Είμαστε πάρα πολύ κατακαιρματισμένοι και σε ό,τι αφορά και με τους, για τους φορείς οι οποίοι είναι διαφορετικού μεγέθους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή και ελελογισμένη διαδικασία μετάβασης σε μια νέα τεχνολογία και σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των φορέων ώστε να μπορούν να επενδύσουν καλύτερα και περισσότερο. Αυτό χρειάζεται μια οικονομική ρύθμιση η οποία να είναι σταθερή και δίνει τα μέσα δράσης με αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη, όπως λέει και η Μπερέκ, την πολυμορφία των εθνικών καταστάσεων και να ακολουθήσουμε το δρόμο της συνεργασίας, την ε, χρήση της νομολογίας που έχει, επί, έχει της κατά νομολογίας που έχει εδρεωθεί και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας. Μια συνολική λοιπόν μεταρρύθμιση θα μπορέσει να γίνει όπως είπε η Κομισιόν και η μπερέκαλα αλλά είναι πολύ πρόημο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πρόωρο να προχωρήσουμε για κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αφαιθούν να γίνουν με μια μεταβατική μεταρρύθμιση. Τα εργαλεία της ρύθμισης, η απλοποίηση της αγοράς, η χρήση, εάν είναι πιο απαραίτητο, μια συμμετρικής ρύθμισης. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία αναφέρονται και από την Κομισιόν και την ΠΕΡΕΚ και όλες αυτές οι προτάσεις μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες. Αν η Κομισιόν λοιπόν θέλει να προχωρήσει για το διαβατήριο του φάσματος και την ουδετερότητα του δικτύου, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην εφαρμογή της ρύθμισης. Και αυτά που είπε ο κύριος Κρότσμαν εξ ονόματος της κυρίας Βαλεάν, αν θέλουμε, αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα, θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα να λειτουργήσει αυτή η συνεκτικότητα. Για να γίνουν λοιπόν όλα αυτά δυνατά δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να αλλάξουμε το σύνολο του συστήματος όπως είπε η Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνεκτικότητα και να διευκολύνουμε αυτή τη συνεργασία η οποία ήδη έχει προχωρήσει σημαντικά μεταξύ της Κομισιόν και της Μπέρεκ. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την όλη προβληματική του διαβατηρίου. Υπάρχει ένα θέμα που η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει απάντηση. Αν έχει κανείς ένα διαβατήριο για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε μια χώρα, τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο φορέας δοσιδοκίας σε περίπτωση κάποιας εμπορικής διαφοράς. Είναι η χώρα η οποία έχει εκδώσει το διαβατήριο, είναι η χώρα που είναι εγκατεστημένος ο φορέας θα πρέπει να υπενθυμίσω την αρχή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες που δίνει διαφορετικά δικαιώματα από ό,τι οδηγία για την εγκατάσταση. Εγώ θα θεωρούσα πάρα πολύ χρησιμό να υπάρξει μια απλοποίηση, αλλά προσοχή, θα πρέπει να ξέρουμε ποιε είναι οι συνέπειε που θα προκύψουν και αν υπάρχουν συνέπειε σε κοινωνικό επίπεδο, χρειάζεται μια μελέτη αντικτύπου, όπως συνιστάται και από το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για, το λεγόμενο, για τη λεγόμενη αποδεσμοποίηση για την οποία αναφέραμε, το unbundling, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και στην ε, ρύθμιση ένα σημαντικό αποτρεπτικό εργαλείο για να αποφύγουμε προβλήματα. Παραμένει λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο είναι στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Σε, στο επίπεδο αυτό θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς για την ανοχή σας, για το χρόνο που μου δώσατε για αυτή τη συζήτηση που είναι σίγουρα πολύ θετική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Κατρίν, ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερος ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους δύο <coughs> καλεσμένους μας από την πλευρά του Μπέρεκ. 9 Ιουλίου, όπως είπα και προηγουμένως, θα συζητηθεί ε, το προσχέδιο της έκθεσης που θα είναι έτοιμο, θα ετοιμάσει η Κατρίν Τροτμάν. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Είναι ε, πάντα για θέματα πληροφορικής. Αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Τοζενόφσκι. Ναι, παρακαλώ πολύ οι αποχαιρετισμοί να γίνουν διακριτικά μέσα στην αίθουσα. Ε, Έχουμε ενώπιον μας τα θέματα αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Έχουν εγκριθεί όλα αυτά από την Επιτροπή Ήτρε το Νοέμβριο. Μετά όμως παρενέβησαν κάποιες αλλαγές ιδίω στη χρηματοδότηση που αφορά το πρόγραμμα αυτό, υπήρξε μια περικοπή από 9,2 δισεκατομμύρια σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και όλη η έκθεση πρέπει να αναθεωρηθεί. Πήραμε μια νέα πρόταση από την Κομισιόν και με την περικοπή αυτή υπήρξαν και ουσιαστικές αλλαγές περιεχομένου και οφείλονται όλα αυτά στο γεγονός ότι το σημείο εστίασης έχει μεταφερθεί στη συστημικού χαρακτήρα υπηρεσίες και το ευρυζωνικό φάσμα έχει πάρει λιγότερη σημασία από ό,τι ήταν το Νοέμβριο όταν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει και νέες ιδέες, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατανομή των ψηφιακών υπηρεσιών με τις συζητήσεις για τη διευκόλυνση Connecting Europe συνδέοντας την Ευρώπη φτάνουμε πια σε ένα χρονικό σημείο που υπάρχει μια πίεση πάνω μας. Και θα ήθελα να εκφράσω τις ε, ευχαριστίες μου για τη συνεργασία που με επιφύλαξαν όλοι οι σκιώδεις συζητητές, γιατί παρά την πίεση χρόνου εμείς αγωνιστήκαμε να μπορέσουμε να βρούμε μία σύγκληση, μια συμβιβαστική λύση σε πολλά θέματα, που θα ήταν ως το δυνατόν ευρύτερη επί τη βάση του κειμένου που ήταν αντικείμενο συζήτηση τον προηγούμενο Νοέμβρη. Προσπάθησα να εξεύρω μία συνένεση όσο το δυνατόν ευρύτερη μεταξύ των σκιών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο στην Επιτροπή Ήτρε πριν από τις χθερινές διακοπές. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δώσουμε εγκαίρως την έκθεση αυτή προς την Ολομέλεια. Η προσπάθειά μας λοιπόν ήταν έντονη και το εκτιμώ αυτό ιδιαίτερα. Το πρόβλημα που βλέπω και εδώ θέλω να σταθώ και να ρωτήσω την Κομισιόν, είναι ότι έχουν παραμείνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την κατανομή αυτό του δισεκατομμύριου ευρώ μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών και των ευρυζωνικών θεμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το δισεκατομμύριο και πώς θα το αντιμετωπίσει η έκθεσή μας πώς θα το ευθυγραμμίσουμε με τα θέματα που έχουμε ήδη αποφασίσει στο παρελθόν. Θα πρέπει να ξέρουμε επίσης από την Κομισιόν αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να αντιμετωπιστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τα ε, μεμονωμένα σχέδια ψηφιακών υπηρεσιών. Γιατί έτσι έγινε η κατανομή των κονδυλίων για μεμονωμένα σχέδια. Πού να βάλουμε την Ευρωπαϊκή και πώς να εξασφαλίσουμε και πιο εύκαμπτο πλαίσιο διαπραγματεύσεων στον τριμερή διάλογο, ο οποίος θα γίνει μετά από το καλοκαίρι. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η επίηση χρόνου, η οποία είναι ζωτική, σημαντική για μας. Και εγώ θέλω να διατηρήσω το χρονικό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα που έχει θεσπιστεί, να το τηρήσω. Γι' αυτό Θα ήθελα να μπορέσω να σας δώσω τις τροπολογίες αφού συμφωνηθούν από τους κοιόδης συζητητές το ταχύτερο δυνατό τις συμβαστικές τροπολογίες. Όταν λοιπόν περατωθεί αυτή η διαδικασία θα ήθελα να εξασφαλίσω την ευρύτερη δυνατή συνένεση σε επίπεδο συμβιβασμού μεταξύ όλων των σχεδόν ισογητών Προσβλέπουμε λοιπόν στον τριμερή διάλογο. όπου θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα αυτά και με το Συμβούλιο και όπου θα πρέπει να, συμβεί, να βρεθούμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Γι' αυτό σας ζητώ να έχω όλες τις τροπολογίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες, απλώς θέλω να τονίσω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τους σκιώδεις εισηγητές. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή να παραμείνουμε στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος. Γι' αυτό σας ζητώ να καταθέσετε όλες τις τροπολογίες σας αυτή τη βδομάδα. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς αποδεκτούς από όλες τις πολιτικές ομάδες και έτσι να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι πράγματι πολύ πιεστικό. Δύο ερωτήματα τώρα προς την Κομισιόν. Τι πιστεύετε για το θέμα της κατανομής των πόρων μεταξύ των διαφόρων κεφαλαίων. Αυτό θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα για το έργο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Έχουμε εντωμεταξύ τον δόκτωρα Βιόλα, ο οποίος ήρθε για να μιλήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ξεκινήσουμε με τον Σνέφο Όκμαρ, κάνοντας το γύρο των ε, σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Ιδιαιτέρως εκτιμώ όχι μονάχα την παρουσία του, αλλά και ε, τον δρόμο που έχουμε διανύσει με αυτή τη δύσκολη διαδικασία ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες ε, των, ε, του MFF. Τα ζητήματα είναι δύο ειδών. Το ένα είναι τα κριτήρια και οι στόχοι και το δεύτερο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση. Πώς μπορούμε δηλαδή να βρούμε τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτά που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Όσον αφορά τους στόχους και κριτήρια, σε αυτό το σκέλος δεν έχει αλλάξει κάτι. Άλλαξε ο προϋπολογισμός βέβαια. Αλλά δεν έχει αλλάξει η πραγματικότητα ούτε το συνολικό πλαίσιο. Δεν συμφωνώ απολύτως με την Κομισιόν στην αναθεωρημένη πρόταση, εκεί που λέει ότι ε, δεν είναι πολύ εύκολο ε, στην, ε, στην, ε, στην Ήπεθρο να υπάρξουν μεγάλες ταχύτητες. Όχι, εγώ λέω το αντίθετο, ότι πρέπει η ψηφιακή πραγματικότητα να είναι εντελώς διαφορετική πλέον. Γιατί αν πούμε εξ αρχής ότι οι ταχύτητες για το 2013 είναι αρκετές και για το 20, τότε είναι σαν να δηλώνουμε ότι το 2020 θα υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, ψηφιακό χάσμα και ότι οι οικονομίες της υπεθρού δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όπως είπε και ο εισηγητής άλλωστε, είναι σημαντικό να επανυποβάλουμε τις ε, ε, τροπολογίες ε, τις οποίες είχε στηρίξει η Επιτροπή στην τελευταία ψηφοφορία. Τώρα, τι θα γίνει με τα οικονομικά. Αν δούμε τη συνολική εικόνα, 9 δις ευρώ είναι βεβαίως πολύ περισσότερο από τι 1 δις. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο μιλητής, είναι 9 φορές περισσότερα. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο εύρος των ε, επενδύσεων που πρέπει να γίνουν, και αυτά τα εννέα δις δεν είναι πολλά, πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις επενδύσεις. Και ένας τρόπος κινητοποίησης των σωστών επενδύσεων είναι ε, να είναι κανείς σαφής όσον αφορά τους στόχους και τα κριτήρια. Το template πρέπει να είναι για το μέλλον και για τις κινήσεις μας του μέλλοντος, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, σαφές έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους και επενδύσεις. Αυτό είναι σημαντικό και για την Κομισιόν αλλά και για τη συνολική συζήτηση. Και βεβαίως να πω ότι στηρίζω ε, ιδιαιτέρως την ε, τοποθέτηση του ε, εισηγητού. Και ξαναλέω ότι μπορεί να άλλαξαν οι χρηματοδοτικές μας ικανότητες, αλλά δεν έχει αλλάξει ο κόσμος. Επομένως, ξέρουμε ποιες είναι οι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να στηριχτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς πρέπει να στηριχτούν με άλλο τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε ορθολογιστές, θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε αυτή την ορθολογική, πληνμένα αποφασιστική γραμμή που προτείνει ο εισηγητής. Αυτή τη γραμμή να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε Όκμαρ. Ε, η κυρία Τροθμάν, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία που πραγματικά συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία με τους ε, σκιώδεις και τον ευχαριστώ που μας άκουσε. Ε, σε ένα βαθμό συμμερίζομαι κι εγώ αυτά τα θέματα γιατί και εμάς μας απογοήτευσε ο τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετωπίσαμε το θέμα των ψηφιακών δικτύων, πώς θα αντιμετώπισαν αυτά τα θέματα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, που δεν αναγνώρισαν αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος, ότι αυτά τα δίκτυα είναι καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να τα συζητήσουμε όπως ε, έχει γίνει αγαπητέ συνάδελφοι. Να συζητήσουμε λοιπόν για τα δισεκατομμύρια που μένουν και έχουν ε, καταναμηθεί στα ψηφιακά δίκτυα. Υπάρχει το ζήτημα των υποδομών. Εφόσον έχουμε μόνο ένα δις πλέον, θα μιλήσουμε για τις υπηρεσίες, αλλά δεν θέλω το Κοινοβούλιο να μείνει έξω από τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Εάν αυτό το πρόγραμμα δεν μας επιτρέπει να συζητήσουμε τα δίκτυα και αφήσουμε τη χρηματοδότηση ε, στον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα, είναι σημαντικό να μην τεθεί κατά μέρο το κοινοβούλιο. Αυτό ήθελα να πω, γιατί έχουμε και εμείς να πούμε κάτι σε αυτή τη συζήτηση. Αν δείτε και την συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Και απογοητεύτηκα και εγώ όταν είχαμε την ε, συνεδρίαση για τη συνάντηση με την κυρία Κρούς και είχαμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν θέλω να κάνω προσωπική επίθεση, αλλά μας εξήγησε ότι ε, τα ποσοστά δανειοδότησης για ε, τις υποδομές ήταν πιο αυξημένα, ήταν υψηλότερα σε αυτή την περίπτωση των δικτύων τηλεπικοινωνίας σε σχέση με την ενέργεια για τις μεταφορές. Γιατί θεωρούνται πιο ρηψοκίνδυνα, αν θέλετε. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε είπε ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη έρευνα ή μάλλον να βρούμε περισσότερες δημόσιες εγγυήσεις. Όμως ε, εδώ δεν μπορούμε να ζητήσουμε επενδύσεις γιατί δεν μειώνονται, δεν αφαιρούνται από τον ε, υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματος και ούτε μπορούν να δοθούν τέτοια δημόσια εγγύα. Δεν έχουμε λοιπόν ξεφύγει από τα δύσκολα σε ό,τι αφορά τι επενδύσεις στα κράτη-μέλη για αυτά τα δίκτυα. Και αν δείτε και πώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιλέγει τα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσει, θα δανειοδοτήσει, στα ε, προγράμματα των μεταφορών αφορούν αυτοκινητοδρόμους. Δεν είναι τα προγράμματα που στη διαδικασία της συναπόφασης ε, θεωρούνταν ως ε, προγράμματα προτεραιότητας που να αφορούν δηλαδή την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο και στο διαδίκτυο. Πρέπει να δούμε με ποιου όρου υπάρχει αυτή και αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών, πληθυσμιακή διάσταση, γεωγραφική διάσταση. Πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε ε, μια ισότητα βεβαίω για όλα τα κρατημέλη, αλλά θα πρέπει να σταθούμε και από αυτή την ανάπτυξη που επιθυμούμε. Και Σήμερα πρέπει να μεταφέρουμε ένα μήνυμα που να το ακούσει και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις, ιδίως για το 5-3-β, ε, για να υπάρξει ένας δημοκρατικός προσανατολισμός στις επιλογές που γίνονται. Αυτά για τις υπηρεσίες. Ε, σίγουρα η προσέγγιση είναι πολύ σωστή, όμως έχουμε λιγότερα μέσα. Επομένω, καλό θα ήταν να επιλέγουμε καλύτερα τα προγράμματα. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Γιατί έχουμε, αν έχουμε αυτό το ένα δις μόνο, αυτό γρήγορα θα απορροφηθεί. Και ανησυχία όλων μας είναι να καταφέρουμε να είμαστε ως τον πιο αποτελεσματικοί με αυτό το μειωμένο κονδύλι. Συγχαίρω τον συνάδελφο εισηγητή. Θα εξεύρουμε ένα συμβιβασμό γιατί πράγματι πρέπει να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου με έναν συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Όλοι συμμεριζόμαστε αυτό τον στόχο της αποδοτικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής, ε, συγγνώμη, ο Σκιώδης, της άλλης, ο κύριος Κράτσμαν έχει το λόγο. Μερσή, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, έχω εκφράσει ήδη την άποψή μου στο παρελθόν για το θέμα αυτό, αλλά μπορώ να τα επαναλάβω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η πρόταση αυτή, γιατί συμφωνώ με την ιδέα να εστιάσουμε τα περιορισμένα κονδύλια στα κέρια σχέδια και ιδίως αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Για το θέμα τώρα των ευρωζωνικών υπηρεσιών απαιτείται μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών. Από τα 9 δισεκατομμύρια έχουμε πέσει στο 1, το οποίο είναι μονάχα σταγόνα εν το ωκεανό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα κονδύλια. Η απόφαση φυσικά είναι κάτι που θα γίνει από τα κράτη-μέλη και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει νόημα να το συζητήσουμε περισσότερο. Ερχόμαστε τώρα στο άλλο θέμα που είναι η υποδομή για τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες. Υπάρχει μια πλειάδα από προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν από το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Η ηλεκτρονική υπογραφή, οι ηλεκτρονικές προμήθειες και η ηλεκτρονική υγεία μας δίνουν τεράστιες δυνατότητες στην αγορά μας. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα νομοθετικής ρύθμισης τα οποία πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να αναφέρω επίσης και την, τον ρόλο των ηλεκτρο, ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τα εθνικά μητρώα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Εδώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει νέα μέσα τα οποία μπορούν να δώσουν προσθέμενη αξία και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες της Ευρώπης το πρόγραμμα Ευρωπαίνα δεν πρέπει <clears throat> να περικοπεί και ευτυχώς δεν έχει υποστεί μεγάλες περικοπές από την μείωση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της, του σχεδιασμού και επίσης πρέπει να αναζητήσουμε για το πρόγραμμα αυτό και νέες πηγές χρηματοδότησης όσο και δύσκολο να είναι μέσα στην τωρινή οικονομική κρίση. Και τώρα για το ασφαλέστερο ίντερνετ υπάρχουν ορισμένα μέτρα τα οποία μπορεί να θεωρούνται αφισβητήσιμα από ορισμένου συναδέλφου, όπω παραδείγματο το σβήσιμο των σελίδων που είναι επιλήψιμε. Είναι απαραίτητο όμω να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Έχουν επενεθεί οι αντίστοιχε πρωτοβουλίε στη Γερμανία για την προστασία των ανηλίκων και το μεγαλύτερο ρόλο των γονέων τους. Και με το Connecting ε, Europe υπάρχει και μια υποδομή η οποία προβλέπεται να δημιουργηθεί για το διαδίκτυο το αν αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα ε, και η ανάγκη να έχουμε περισσότερες εκστατείες για την ασφάλεια του διαδικτύου είναι κάτι το οποίο τονίζεται και στο κείμενο μας. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε πάντα να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και εδώ μιλώ και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και να μπορέσουμε να αποκομίσουμε και τη δική τους υποστήριξη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Επομένως εδώ θα πρέπει να είναι προσεκτική η Κομισιόν με τον τρόπο που θα κατανείμει τα κονδύλια για τις ευζωνικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Είναι και ιδιαίτερα φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, αλλά με τη συνεργασία όλων θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. E- Ευχαριστώ πολύ. Ε- το, λόγο έχει η συνάδελφος ε, Ντότερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση για, την, για το αθεωρημένο κείμενο της ε, Κομισιόν και από την πλευρά των Πρασίνων είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν όσο γίνεται περισσότερα από τα πράγματα τα οποία πέρσι σχεδόν ομόφωνα αποφασίσαμε. Ε, έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους λοιπόν ε, για την ευρυζωνικότητα και πιο σαφή κριτήρια και στόχους για κοινού συμφέροντος ε, στοιχεία θα ήθελα να πω ότι εξακολουθώ να στηρίζω τις, τη δημιουργία υποδομών έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα σε ενωσιακό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το ψηφιακό χάσμα το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι ήδη μεγάλο. Ε, πρέπει να πω ότι από την αρχή είμαστε λίγο διστακτικοί να βάλουμε και τις υπηρεσίες σε ένα κείμενο που πολύ μιλάει για υποδομές. Ε, είναι λίγο ξένο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές το έχουμε δει να συζητιέται και μάλιστα και λίγο πριν σήμερα το συζητήσαμε ε, όσον αφορά ε, στα πλαίσια μάλλον του θέματος ηλεκτρονικής ε, ταυτοποίησης και της υπηρεσίας εμπιστοσύνης. Πρέπει να το δει κανείς πιο συνολικά. Με μεγάλη χαρά ακούω τον εισηγητή να αναφέρεται σε προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό, ας πούμε. Μα ικανοποιεί αυτό, είναι ένα προχωρημένο πολιτιστικό πρόγραμμα. Και πραγματικά εγώ σαν πολίτης, σαν νέος πολίτης της Ευρώπης, κάτι τέτοιο περιμένω να κάνει η Ευρώπη για μένα. Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάτι πριν το 1995 Πολλές κοινωνικές αλλαγές ε, ε, έλαβαν χώρα όμως πριν το 1995, τις οποίες πρέπει να γνωρίζω. Οι οικονομικές, κοινωνικές μάχες, αγώνες στα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία ε, άρρηκτα συνδεδεμένα με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και επομένως πρέπει να έχουμε και προγράμματα σαν το Ευρωπαϊκό γιατί είναι ένας τρόπος διασύνδεσης των πολιτών και νομίζω ότι και πολλοί άλλοι νέοι ε, μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα ε, θετικά ε, στοιχεία από τέτοιου είδους προγράμματα ιστορίας και πολιτισμού. Πολύ ωραία. Άλλοι συνάδελφοι, τελείωσε ο γύρος των σκιωδών. Άλλοι συνάδελφοι, συνάδελφος, η κυρία Φόη. Ευχαριστώ πολύ και, ε, τον εισηγητή ε, και τους σκιώδεις που αναφέρθηκαν σε κάποιες τροποποίησεις που έχουν ε, λάβει χώρα. Έχω ένα ζήτημα το οποίο να θέσω, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Κάποιες λέξεις οι οποίες διαγράφησαν στην σελίδα 38 όσον αφορά την ασφάλεια κυρίως σε σχέση με οργανώσεις, ε, γραμμές βοήθειας, helplines και ειδικές γραμμές hotlines. Child sex continent. Ιδίως ε, ε, περίεργου περιεχομένου που βρίσκονται στο ίντερνετ ε, υπάρχουν ε, μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται σε 30 χώρες. Ε, καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτού του είδους η εγκληματικότητα η οποία προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε μια νέα διατύπωση στη σελίδα 26 όπου γίνεται λόγος για πλατφόρμες διασυνοριακές, διακρατικές ε, πλατφόρμες. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ε, συγκεκριμένοι να πούμε ότι η χρηματοδότηση θα εξακολουθήσει να υπάρξει σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορούν ε, όταν έχουν βρει κάποιο περίεργο περιεχόμενο επιγραμμικά online να μπορούν σε συνεργασία με την αστυνομία να το βγάζουν, να γίνεται offline. Ελπίζω να μπορέσω να συνεργαστώ με τον ε, εισηγητή ε, και τον, τους σκιώδες έτσι ώστε να βρεθεί μια διατύπωση ε, βάσει της οποίας να εξακολουθεί να υπάρχει χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο για τέτοιου είδους οργανώσεις. Υπάρχει η δήλωση υπ. 3 για το ίδιο θέμα. Όσοι δεν την έχουν υπογράψει παρακαλώ να το κάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί οι κίνδυνοι που κρύβονται σε αυτού του είδους τις σελίδες είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Ευχαριστώ πολύ, Ο συνάδελφο Οντί έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Οντί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι μεταξύ των κοινοβουλευτικών οι οποίοι απογοητεύτηκαν πάρα πολύ από το μεγάλο αλογοπάζαρο που έκαναν οι, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το Φεβρουάριο <clears throat> και όπου τα διευρωπαϊκά δίκτυα έπεσαν θύματα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, ο οποίος έχει γίνει ειδικό σε όλα αυτά τα θέματα, ο οποίος έχει εργαστεί πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε για τους επιδιωκόμενους στόχους. Βέβαια υπήρξε το πρόβλημα της χρηματοδότησης αυτά που ζήτησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν έχουν γίνει πραγματικότητα, ζητήσαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβεί σε μία μελέτη για τις γενικές δυνατότητες χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εμπλέκοντας τις περιφέρειες, τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα, εγγυήσεις, ε, επιδοτήσεις κτλ. Δηλαδή τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια καινοτόμα διαδικασία επενδύσεων και είδαμε ότι ένα από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τομέα των, των τηλεπικοινωνιών, είναι να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε όχι τις κερδοφόρες επενδύσεις που θα γίνουν ούτως ή άλλως, ούτε τις επενδύσεις που δεν είναι κερδοφόρες και που δεν θα γίνουν ποτέ, αλλά τις ε, επενδύσεις στην ΦΕΑ περιοχή όπου χρειάζεται και κάποια βοήθεια από το δημόσιο τομέα. Αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εγώ καταλαβαίνω τους ηγέτες της ε, ΕΤΕ που θέλουν να διατηρήσουν την ε, <clears throat> βαθμολογία τριπλού α και επομένως προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν. Αλλά υπάρχουν οι ειδικοί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι ειδικοί στην ε, χρηματοπιστωτική μηχανική και θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ίδιους πόρους για όλα αυτά και στο έγγραφο αυτό μιλάμε για την αξιολόγηση στη μέση του δρόμου. Εγώ σκέφτομαι περισσότερο μια αναθεώρηση πολιτικού χαρακτήρα, γιατί αυτά τα οποία ζητούμε, και εδώ πρέπει να καταλάβουμε τις χρηματοδοτικές δυσκολίες που έχουν τα κρατημέλη δεν μπορούμε να μην δεχτούμε το 1 δισεκατομμύριο που μας δίνεται αντί για εννέα αλλά ας το δεχτούμε μονάχα προσωρινά. Ας περιλαμβάνει ο κανονισμός αυτός ότι μια ρήτρα, όχι αναθεώρησης, όχι ενδιάμεσης αναθεώρησης, αλλά μιας πραγματικής πολιτικής αναθεώρησης, ας, πρέπει το Ευρωπαϊκό, ας αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει το γεγονός ότι θα έχουμε μια νέα κομισιόν, ένα νέο πρόεδρο, του Συμβουλίου νέες εκλογές, ίσως ότι θα φύγει το, Ευρωπαϊ... το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν πολλά πολιτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αλλάξουν βάθρων το επίπεδο επενδύσεων στα διευρωπαϊκά δίκτυα και ιδίως στα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη από τον ιδιωτικό τομέα στα εγχειρήματα αυτά αν δεν υπάρχει επένδυση του δημοσίου τομέα. Είναι καλή λοιπόν η επιχειρηματολογία, αλλά πρέπει να την τροποποιήσουμε για να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει τη δυνατότητα ελπίδας για επενδύσεις σε αυτές τις φαιές περιοχές όπου δεν θα υπάρξει επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς τη βοήθεια του δημοσίου. Η συνάδελφος ζήτησε να παρέμβει εκ νέου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για τη δευτερολογία. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε και τη συζήτηση μεταξύ των σκιωδών. Αλλά να πω κάτι. Ε, ε, εγώ σαν ε, νέα χρήστης των δικτύων υπάρχει κάτι που μου δημιουργεί ανασφάλεια. Μην λησμονείτε ότι αυτοί οι, οποίοι, οι οργανισμοί οι οποίοι παίρνουν χρήματα από το Safer Internet έχουν ε, συμφέρον να συνεχίσουν την ε, παρουσίασή τους. Δηλαδή κάνουν διάφορες περίεργες κινήσεις όπως καταχρηστική ε, λογοκρισία ή καταχρηστικό κλείσιμο κάποιων σελίδων, φιλτράρουν κτλ. Γιατί αυτό, και αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή οι άλλοι αποφασίζουν σε μια πλατφόρμα τι μπορεί να πει ο καθένας και με, ποιος, ε, με ποιες συνθήκες, με ποιες προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό είτε ε, για το καλό των πολιτών, είτε ε, καλό για τους πολίτες ή για τους χρήστες. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να το διεκδικήσει και ο δημόσιος τομέας. Φαίνεται ότι εκεί μυστικά και κρυφά έχουν ε, και διάφορες δομές ε, βοήθειας business to business ε, για αυτές τις περιπτώσεις έτσι. Νομίζω ότι οι 25.000 υπάλληλοι της Κομισιόν θα έπρεπε να είχαν ήδη καταλάβει ότι αυτού του είδους ε, η παρέμβαση ούτε βοηθάει, ούτε είναι αποτελεσματική, ούτε ε, έρει τους ε, κινδύνους. Στην Γερμανία έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση που κράτησε και δύο χρόνια για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτού του είδους προβλήματα, πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ας πούμε, της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και ε, τελικά αποφάσισαν ε, ότι οι ίδιοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία των εικόνων παιδικής πορνογραφίας θα πρέπει να καταδικάζονται. Ε, αυτοί που παίρνουν χρήματα από τις δομές για πιο ασφαλές διαδίκτυο ε, τελικά δεν νομίζω ότι κάνουν και πολλά καλά πράγματα. Το να συνεχίσει αυτό το safer internet ε, δεν νομίζω ότι κάνει καλό σε κανέναν. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτού του είδους οι παρεμβάσεις ε, δεν είναι πολύ... Ναι, θέλετε να σας δώσω το λόγο, φαντάζομαι, στην αλφεφόρντ Κοιτάξτε, Νομίζω ότι έχουμε το χρόνο σήμερα και επομένως θα δώσουμε την δυνατότητα ε, για δευτερολογία και στην συνάδελφο Φόρτ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας καλέσω να δείτε στην δική μου περιφέρεια για να δείτε τον οργανισμό που ε, καταπολεμά αυτή την ε, κατάχρηση στο διαδίκτυο και να δείτε το έργο που επιτελούν. Μην λέτε ότι οποιοδήποτε έχει χρηματοδοτηθεί από αυτό το πρόγραμμα δεν κάνει καλή δουλειά. Sì, prego collega Kreuzmann. Το υποστηρίζω αυτό απόλυτα. Δεν πρόκειται για να Κρίνουμε κανένα, κύριε Άντερς Δότερ. Κανείς δεν το θέλει και το έχουμε συζητήσει αυτό στη Γερμανία. Αλλά θέλουμε, ξέρουμε προγράμματα όπως το ClickSafe, που μπορεί κανείς να προστατεύσει τα παιδιά από την παιδική πορνογραφία, από τις ε, ακροδεξιές οργανώσεις κτλ. Και, και να προστατεύσει έτσι τους ανηλίκους. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε με τους παρόχους ώστε να μπορούν να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση για την προστασία των νέων. Δεν είναι λογοκρισία του ίντερνετ. Γι' αυτό υποστηρίζω λοιπόν δεν πρέπει να το συγχαίρεται αυτό με την ε, λογοκρισία. Είμαστε όλοι κατά της λογοκρισίας. Πολλές φορές όμως οι φορείς και οι πάροχοι δέχονται τις ενέργειες αυτές που γίνονται για την προστασία των περών. Δεν μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε στο ίδιο καλάτι. Μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε την προστασία των νέων και αυτό είναι σίγουρα προς το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές ε, τις αποσαφηνήσεις, διευκρινήσεις σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Πριν ε, δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, ε, να πω και εγώ δύο λόγια στο θέμα το οποίο έθιξαν πολλοί συνάδελφοι και που αφορά το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν επιπλέον πόροι. Γιατί και εγώ λυπούμε, λυπούμε που όπως και άλλοι συνάδελφοι που ε, η χρηματοδότηση δεν είναι ικανοποιητική, δεν είναι αρκετή. Λυπούμε γιατί φαίνεται ότι τα διάφορα κράτη-μέλη και η Κομισιόν δεν καταλαβαίνουν ε, πόσο ε, σημαντικά είναι τα θέματα αυτά για την οικονομική και λυπή ανάπτυξη των χωρών και ελπίζω ότι στη ρήτρα αναθεώρησης θα υπάρχει κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Ένας πολύ αυστηρός προπολογισμό για τα επόμενα χρόνια μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και να ανασχέσει την ανάπτυξη. Ε, να πω το εξή λοιπόν και ελπίζω ότι θα, φανεί, θα διαφανεί αυτό και στις τροπολογίες. Εμείς ε, συχνά έχουμε διάφορα προγράμματα όπως το COSME. Ε, έχουμε λοιπόν ενεργοποιήσει πολλά προγράμματα για επενδύσεις αλλά βράχοι πρόθεσμες για μικρές περιόδους, βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες λοιπόν. Έχουμε και διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη, ανέφερα ήδη και το πρόγραμμα COSME, έτσι ώστε να έχουμε έστω και μικρή, αλλά πάντως κάποια χρηματοδότηση για τη δημιουργία λοιπόν υποδομών, αλλά και για αυτές τις υποδομές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε αυτές τις ε, προϋποθέσεις ε, οι οποίες θα κινητοποιήσουν, θα κινητοποιήσουν ε, επενδύσεις μέσω και μακροπρόθεσμες. Πώς μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κλίμα τέτοιο, ένα θετικό κλίμα έτσι ώστε και από τον ιδιωτικό τομέα ε, να υπάρξουν επενδύσεις σε πιο μακρόθωρες ε, και επίσης ε, με μία επιστροφή που δεν θα είναι σύντομη, θα είναι μία απόσβεση η οποία θα έρθει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ελπίζω λοιπόν μέσω κάποιας τροπολογίας να υπενθυμίσουμε και αυτό που είπε και ο εισηγητής προηγουμένως, δηλαδή ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο Η επόμενη Τρίτη, 22 του μηνός, είναι η ημερομηνία. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ακούσαμε πολλά και διάφορα. Θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή, τον κύριο Διόλα. Ε, ε, πάντα είναι καλοδεχούμενος στην Επιτροπή μας ε, και θα ήθελα αν είναι δυνατόν να απαντήσει στα σχόλια και στα ερωτήματα τα οποία ακούστηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να εδώ στην Επιτροπή σας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω οι ζητητοί και οι συνεισηγητές, οι σκιώδεις, για τις προσπάθειές τους. Θέλουν να υπάρξει έκθεση της Ήτρε πριν από το καλοκαίρι και να σταλεί στο Συμβούλιο. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να κλείσει αυτός ο νομοθετικός φάκελος το συντομότερο δυνατόν για να μπει και αυτή η πρόταση στο τρένο του Connecting Europe. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Πρέπει να αλλάξουμε το σημείο εστίαση και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της σημαντική μείωση του υπερπολογισμού. Θα προσπαθήσω να δώσω περαιτέρω διευκρινήσεις για τα όσα έχουν υποθεί σήμερα για να εξετάσετε και εσείς την πρότασή μας. Πρώτον, θα ήθελα να εξηγήσω πώς ε, σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του προϋπολογισμού. Έχουμε μόνο ένα δις. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Στην... Με την πρότασή μας θα επικεντρωθούμε στις υπηρεσίες και λιγότερο στις ε, υποδομές. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει η κατανομή. Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ευελιξία, αλλά για τις υποδομές ε, υπολογίζουμε να δοθεί κάτω από το 20% του συνολικού κονδυλίου. Βεβαίως δεν έχει κλείσει οριστικά αυτό το ποσοστό αλλά θα είναι μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως να σταματήσουμε κάπου στη μέση, στα 150. Αυτά έχουμε κατά νου για την στήριξη των υποδομών και τα υπόλοιπα θα πάνε στις επενδύσεις, στις υπηρεσίες, συγγνώμη, το 85% περίπου του προγράμματος. Τι μπορούμε να κάνουμε με τα χρήματα που θα κατανομηθούν στις υποδομές να διευκρινίσω το εξή. Θέλουμε κι εμείς να υπάρχει δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη. Αν δεν έχει διατυπωθεί σωστά, να το διευκρινίσουμε. Και θα ήταν περίεργο κιόλας να μην θέλουμε αυτές τις ταχύτητες για, ε, για την ύπεθρο και τις αγροτικές περιοχές. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης περισσότερο, όχι στήριξη του προγράμματος. Γιατί ξέρετε ότι κάτω από 100-150 ε, εκατομμύρια δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για την επένδυση στις υποδομές. Αυτό ήταν το πρώτο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με αυτά τα χρήματα. Είναι περίπλοκη η κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιο σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων να πει θέλω να αγοράσω μια Ferrari και λέει μπορώ να κάνω μια προκαταβολή. Ναι, ένα ευρώ μπορώ να σας δώσω ως προκαταβολή. Βεβαίως και αυτό δεν ε, μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αν η απάντηση είναι ναι, μπορώ να δώσω προκαταβολή, δώστε μου μισό λεπτό, είμαι επιχειρηματίας, κάτι θα κάνω. Τότε ίσω ο πολιτή να περιμένει. Πρέπει όμως να εξετάσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τομέα πληροφορικής να αποτελέσει τομέα προτεραιότητα, Θα ήταν πολύ καλή ε, επιλογή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τότε μπορούμε να εξετάσουμε την βέλτιστη ε, κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων για την στήριξη των επενδύσεων. Τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συμπληρώσουν ε, τι ιδιωτικέ επενδύσεις και έτσι αυτά τα κονδύλια θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, και να συντονίσουν και τις επενδύσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι θέλουμε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, τα κονδύλια των διαφορετικών ταμείων. Δεν τα παρατάμε. Αντιθέτως, ακούσατε και ποια είναι τα δικά μας σχέδια, ότι θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ομογένεια, ομοιογένεια ε, στην εσωτερική αγορά. Και αυτό θα γίνει και μέσω τη βέλτιστης αξιοποίηση των διαθετικών ταμείων. Συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε πώ ε, ε, μπορούν να δράσουν καταλητικά αυτά τα χρήματα. ούτω ώστε οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια και υπάρχουν και κάποιες καινοτόμες ιδέες, τις οποίες θέλουμε να δοκιμάσουμε στο ΣΕΦ. Εκεί θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια με πιο δομημένο τρόπο στις υποδομές με τα ταμεία. Περνώ στις υπηρεσίες. δεν έχουμε προτείνει κατανομή ε, των κονδυλίων μεταξύ των υπηρεσιών που υπάρχουν στον κατάλογο. Για δύο λόγους. Πρώτον, ομολογώ ότι δεν θα υπάρξουν ε, αρκετά κονδύλια για να καλύψουμε όλες ε, τις προτάσεις που έχουμε, όλα τα αιτήματα φορέων που έχουν προτείνει, ποια είναι τα προγράμματά τους, και ποια είναι τα κονδύλια που χρειάζονται. Όποιο και αν είναι το συνολικό ποσό θα είναι περιορισμένο. Και υπάρχουν πολλές και σημαντικές υπηρεσίες. Ε, πολιτισμός, ασφαλές διαδίκτυο, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ανοιχτά δεδομένα, όλα εξαιρετικά σημαντικά. Θέλουμε να δούμε και ποια θα είναι η γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ποια θα είναι η τελική συμβιβαστική λύση. Έτσι έχει η κατάσταση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της έλλειψης πόρων, στη νέα πρόταση έχουμε κάποια κριτήρια για την επιλογή, δηλαδή οι υπηρεσίες θα πρέπει να δουν κατόπιν εξάντλησης ε, των κονδυλίων πρέπει να δουν πώς ακριβώς θα ε, εξεύρουν χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει με εμπορικό τρόπο. απαραίτητος. πρέπει να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για να δούμε κατά πόσο μπορούν να επιβιώσουν μόνες τους, ε, κατά πόσο μπορούν να είναι αυτάρκεις ε, αυτοί οι οργανισμοί. Και αυτό θα είναι κριτήριο κατανομής των κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Βεβαίω και θα υπάρξει κάποια ευελιξία στην κατανομή των πόρων. Θα δούμε το πρώτο πρόγραμμα εργασιών και θα, μετά θα κάνουμε την τελική μας κατανομή. Και πάλι όμως είμαστε απολύτως ανοιχτοί και διατεθειμένοι να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο την πρότασή μας. Κυρία Πρόεδρε, αυτά είναι ο Να σας μεταφέρω και τι μάθαμε από την παρουσίαση που κάναμε στα κράτη-μέλη. Παρουσιάσαμε λοιπόν το αναθεωρημένο πρόγραμμα στην Κορεπέρ και η Προεδρία παρουσίασε έκθεση προόδου ε, στο Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου. Βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές ε, υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών. ευρεία στήριξη από πολλά κρατημέλη, αλλά και σημαντικές αντιδράσεις. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Συμβούλιο. ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υπάρχει πάλι ευρεία στήριξη. Και υπάρχουν και κάποια πιο θεσμικά ζητήματα, ο ρόλος των ομάδων εμπειρογνωμόνων και πώς ε, θα οργανωθεί το δικό τους πρόγραμμα εργασιών. Κλείνω εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. E- σας ευχαριστούμε. Και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις ε, στο εργασίες του Συμβουλίου, αν θα υπάρξει πρόοδος ή όχι. Για να κλείσουμε δίνουμε το λόγο στον κύριο και τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους. Ξέρουμε ότι ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι πολύ λίγα λεφτά και δεν μπορούμε με αυτά τα χρήματα να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε ενώπιόν μας. Συμφωνώ και με τον κύριο Οντί, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης για το μέλλον και να υπογραμμίσουμε τη σημασία όλων αυτών των ε, προγραμμάτων. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε όλα αυτά τα προγράμματα που είναι τόσο σημαντικά για το μέλλον. Και αληθεύει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν και νέες αντιμετωπίσεις για τη χρηματοδότηση στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο θα εγκριθεί, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας. Θα υπάρξουν και άλλα έγγραφα και άλλα, άλλες φάσεις για την εργασία μας. Νομίζω ότι αυτό το ένα δισεκατομμύριο είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να τονίσουμε τις μελλοντικέ κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Θα πρέπει να διασυνδέσουμε όλους τους εμπλεκομένους και ξαναλέω και για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά. Να τονίσω επίσης τις υπηρεσίες που εξασφαλίσουν την ασφάλειά μας. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε φυσικά την λογοκρισία, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα μας επιτρέψει να λύσουμε προβλήματα προστασίας των ανηλίκων κτλ. Εγώ είμαι κομπιουτερά στο επαγγέλμα και θυμάμαι πολλές ε, συνδιασκέψεις όπου θελήσαμε να προστατεύσουμε τους χρήστες από το παράνομο και ε, βλαπτικό περιεχόμενο. Είναι δύσκολα τα προβλήματα αυτά. Είναι πολλά τα αδικήματα που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο γιατί είναι ένας ανοιχτός χώρος. Πρέπει επομένως να δώσουμε και έμφαση στην εκπαίδευση των Χριστών. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειε, απλώ σα λέω ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ όλου του συναδέλφου οι οποίοι με υποστήριξαν γιατί έχουμε πράγματι αυτή την πίεση χρόνου. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, Ολοκληρώνεται η πρωινή μας ε, εργασία, η οποία αφορούσε εξ ολοκλήρου την ε, πληροφορική αυτόν τον τομέα. Ξέρετε ότι δεν ε, έχουμε το θέμα της ενημέρωσης για τον τριμερή διάλογο. Θα ξαναρχίσουμε λοιπόν ε, στις 3 ε, η ώρα. Η συνεδρίασή μας όμως θα λάβει χώρα στην 6Q2 στο κτίριο Γιάννα. Ε, τελειώσαμε πιο νωρίς, έχουμε λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο για μας. Πολύ ωραία, καλό μεσημέρι.